Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύσω την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής μας σήμερα. Πάμε μέσα στο σημείο 1, έγκριση της μέσης διάταξης, την έχετε λάβει. Θα σας πρότεινα μια αλλαγή στο σημείο 8, που είναι η ψηφοφορία για την ελεύθερη συμφωνία με την Τινησία, ε, να αναβληθεί το σημείο αυτό, η ψηφοφορία και το σημείο 10 που είναι προφορική ερώτηση για την οικονομική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικής Αφρικής, τη συμφωνία δηλαδή, να μην κάνουμε συζήτηση, αλλά να ψηφίσουμε κατευθείαν. Ε, διαφωνεί κανείς? Όχι. Ωραία. Με αυτές τις αλλαγές λοιπόν εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και πάμε μέσα στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ξέρετε ποια είναι η πάγια τακτική μας. Εάν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν έχουν κατατεθεί αιτήματα για αλλαγέ των πρακτικών, θεωρούνται αυτά εγκεκριμένα. Σημείο 3 στη μέση τέταξη ανακοινώσει του Προέδρου. Και εδώ θα περιοριστώ στη γνωστή ανακοίνωση ότι μεταδίδεται η συνεδρίασή μας απευθείας και όλοι οι θεατές μας βλέπουν. Λόντρα, Παρίσι, Βουδαπέστη, Λούνεμπεκ, Λισαβόνα και Βιέννη. Είναι γύρω στους 300 κυρία Επίτροπη για να ξέρετε που παρακολουθούν τις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής μας απευθείας. Έχετε λάβει και ένα κατάλογο αλληλογραφίας. Αν θέλετε να κοιτάξετε τα γράμματα αυτά, η γραμματεία θα σας βοηθήσει. Και έρχομαι μέσα στο σημείο 4. Γι' αυτό αρχίσαμε νωρίτερα σήμερα. Χαίρομαι που καλωσορίζουμε την Επίτροπό μας εδώ, την κυρία Μάλμστρομ. Καλωσορίστε θερμά κύριε Επίτροπε. Μόλις επέστρεψε από τον Ταβούση η κυρία Μάλμστρομ, όπου θα δούμε και τα θέματα της συμφωνίας στο Ναϊρόμπι και ε, αυτό συζητήθηκε και στον Ταβός από ό,τι ξέρω. Γνωρίζετε ότι είχαμε πάει όλοι μαζί στο Ναϊρόμπι 15 με 19 ε, Δεκεμβρίου και παρόλο που η οι προποθέσει από τι οποίε ξεκινήσαμε δεν ήταν πάρα πολύ ευνοϊκέ. τελικά επετεύχθη η συμφωνία σε ό,τι αφορά την απαγόρευση των γεωργικών επιδοτήσεων και κάποιες παραχωρήσεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Γενικώ πάντως και η διαδικασία πρέπει να πω αξιολογείται πάρα πολύ θετικά. Οπότε ορισμένοι που έσπευσαν να ισχυριστούν ότι ε, εξέλιπε ο ΠΟΕ διαψεύστηκαν οι κασάδρε αυτέ Καλή ήταν η εξέλιξη. Τώρα δεν θα σα πω τι έγινε στο Ναϊρόμπι, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε τι διαπραγματεύσει, Η κυρία Μάνσον θα τα κάνει αυτά. Επίτροπο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, Καλή χρονιά σε όλου. Προσβλέπω σε άλλη μια χρονιά της Ναι, όταν συνηθήκαμε πριν τα Χριστούγεννα στην ίδια αυτή αίθουσα. Ήταν ζωφερά τα μηνύματα τα οποία σας έφερα. Υπήρχε βεβαιότητα ως προς το εάν θα έβγαινε έστω και το παραμικρό από το Ναϊρόμπι. Ακόμη και τις δύο πρώτες μέρες όταν πήγαμε στο Ναϊρόμπι επικρατούσε μεγάλη αβεβαιότητα. Ήδη κάποιοι έγραφαν την εκρολογία του ΠΟΕ και τα όρνεα πέτουσαν πάνω από το κέντρο Κενιάτα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν παρά τις ζωφερές εξελίξεις και τις συνθήκες τις χαοτικές που σας περιέγραψα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης καταφέραμε στον ΠΟΕ να μεταστρέψουμε την πορεία και ο ΠΟΕ λοιπόν ε, ζει και βασιλεύει και μπορεί και παίρνει αποφάσεις πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια επετεύχθη συμφωνία στα γεωργικά. Αυτό είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της πλέον του ΠΟΕ. ικανοποιήθηκαν ε, αιτήματα για πρώτη φορά στον γεωργικό τομέα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, να σας πω εν συντομία τι συμφωνήσαμε και μετά θα σας πω και λίγα λόγια για το Νταβός, για το πώς προχώρησαν εκεί οι υπουργοί την υπόθεση. Πετύχαμε συμφωνία για τον ανταγωνισμό των εξαγωγών στον γεωργικό τομέα. Ξέρουμε ότι το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου είναι πολύ ψηλό. Περαμεινόμεθα και περαμεινόμεθα αυτών των συμφερόντων τόσο πολυμερός όσο και διμερός. Έτσι, από τις αρχές Δεκεμβρίου επιδιώξαμε ένα ισόρροπο αποτέλεσμα, όχι μόνο για να καταργηθούν οι επιδοτήσεις, γιατί αυτό ήταν ένα κίνδυνος, αλλά και για να ε, μπει μια ε, τάξη σε άλλα μέτρα που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα τις εξαγωγές. Το διεθνέ εμπόριο επηρεάζεται βεβαίω από τι επιδοτήσει ε, και αυτό αφορά και μερικού γειτονέ μα. Η δήλωση λοιπόν του, η διακήρυξη του Ναϊρόμπι σηματοδοτεί το τέλος αυτής της εποχής καθώς και μέτρο όσον αφορά τη χρήση, την επιδότηση των εξαγωγών, την επιστημική βοήθεια, ε, κάτι το οποίο θα οδηγήσει ένα πολύ πιο δίκαιο περιβάλλον για όλους. Δεσμευτήκαμε επίση στη διακήρυξη να ασχοληθούμε με την ασφάλεια της τροφοθεσίας σε τρόφιμα, τη διατροφική ασφάλεια, η συμφωνία, το λεγόμενο πακέτο Ναϊρόμπι, όπως προείπα, έχει μια συμβολική σημασία, πολύ σημαντική. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Ο ΠΟΕ παραμένει ο χώρος στον οποίο συνάπτονται διεθνείς συμφωνίες για το εμπόριο. Δύο νέα μέλη, το Αφγανιστάν και η Λιβερία, προσθέθηκαν στον ΠΟΕ, κάτι το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ΠΟΕ είναι ελκυστικός ε, προς νέα μέλη. Πέραν όμω το λεγόμενο υπουργικό πακέτο θα θυμόμαστε τον Ναϊρόμπι γιατί καταφέρουμε να συμφωνήσουμε επί πλειομερών συμφωνιών όπως ε, ήταν καταφέραμε να καταργήσουμε δεσμούς για το 10% των παγκοσμίων συλλαγών μιλάμε για ένα 3 εκατομμύριο περίπου δολάρια έτσι λοιπόν ο τομέας της πληροφορικής θα έχει πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τι νέε, εταιρείε, τις μικρές εταιρείε, τι νεοφυεί εταιρείε, οι οποίε θα έχουν φθηνότερη πρόσβαση σε κάποιε από τι διεθνεί αγορέ, με τα τεχνικά του εξαρτήματα. Η ETA εκτιμάται ότι θα κυρωθεί έω τον Ιούλιο και παρακαλώ η Επιτροπή μα να δει το θέμα των συντομότερων δυνατών. Ε, το συζητούσαμε με τον πρόεδρο πριν από λίγο Τώρα, στο Ναϊρόμπι, στι ε, κατρικέ συνεδριάσεις για την Συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σε θέση να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, γεφυρωτικό θα έλεγα. Ε, ήμουν εκεί σε συνεχεί διαπραγματεύσει με τον Επιτροπό Χόμπαν επί 26 ώρε και πρέπει να σα πω ότι καταρθώσαμε να αποκραστήσουμε επικοινωνία, να ρίξουμε γέφυρε όπω λέμε και να καταλήξουμε στην τελική απόφαση. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαμε τη δική σας βεβαίως υποστήριξη εκείνες τις μέρες. Που πηγαίνω από εδώ και πέρα. Στην διακήρυξη του Ναϊρόμπι, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, λέμε ότι φυσικά ε, δίστανται οι απόψεις ακόμη μετά από την Τόχα. Άλλοι προτείνουν μια νέα εντελώς προσέγγιση για νέα ζητήματα. Η συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον ζει η Ντόχα ή όχι δεν ενδιαφέρουσα, διότι έδειξε ότι ο ΠΟΕ είναι έτοιμος να πετύχει αποτελέσματα. Κάποια θέματα της ΔΟΧΑ επανήλθαν, διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει δουλειά εκεί. Θα συνεχίσουμε το έργο αυτό πάνω στην ατζέντα της ΔΟΧΑ. Όμως, χρειάζονται και νέες προσεγγίσεις, νέα βήματα. Υπάρχουν νέα αιτήματα τα οποία φορούν τη νέα παγκόσμια οικονομία. Το εμπόριο είναι από τα λίγα εργαλεία τα οποία τονώνουν τη διεθνή ζήτηση. Είχα τη χαρά να συναντήσω περίπου 30 υπουργού εμπορίου στον Ταβό. Είχαμε άτυπε συζητήσει για το τι θα γίνει μετά το Ναϊρόμπι. Όλοι ήταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα του Ναϊρόμπι και αποφασισμένοι, θα έλεγα, να αξιοποιήσουν την ε, ορμητικότητα αυτή που έχει προκύψει, γιατί υπάρχουν πολλές καλές ιδέες στο τραπέζι και υπάρχει ομοφωνία για τρία ζητήματα. Πρώτον, πρέπει να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε στο Ναϊρόμπι, αυτό για την αξιοπιστία μας. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα εκρεμή ζητήματα στη διακήρυξη του Νερόμπι και τρίτον πρέπει να εξεύρουμε τρόπους να συζητήσουμε τα νέα θέματα, αυτά που προέκυψαν, όχι ως απειλή στο πολυμερές ζήτημα, στο πολυμερές με συγχωρείτε πλαίσιο, αλλά τουλάχιστον να σημειώσουμε πρόοδο, έστω και να δεν συμφωνούν όλοι από την αρχή. Να ξεκινήσουμε με μικρότερες ομάδες, μικρότερα σύνολα, υποσύνολα και μετά να προχωρήσουμε φροντίζοντας βεβαίως οι θέσεις των λιγότερων ανεπτυγμένων χώρων να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη και αυτό φυσικά να μην απειλεί τις καταλληλα διαπραγματευσεις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν προβλεπόμενες ε, συναντήσεις G20 ε, Σανγκάι τον Ιούλιο, έχουμε το ΟΣΑ στο Παρίσι. Είναι ευκαιρίες να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν εννοείται θα συμμετάσχει επικοδομητικά σε όλους αυτούς τους διαλόγους. Χρειαζόμαστε όμως λίγο χρόνο να σκεφτούμε το πού πηγαίνουμε και εννοείται ότι θα είμαστε σε συνόηση με όλους εσάς. Να δούμε δηλαδή πώς ε, τη θετική αυτή ενέργεια που έχει συγκεντρωθεί θα την αξιοποιήσουμε και με την ευκαιρία ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπήθηκε στο Νερόμπι. Ευχαριστώ για το έργο σας. Και σας ε, λέω για μια φορά ότι πρόκειται μόνο για την αρχή. Προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο λοιπόν συνάδελφοι. Ο κύριος Βίγκλερ πρώτος. Και σας θυμίζω ότι χρόνο έχουμε μέχρι τις 3 και 4. Παρακαλώ σύντομες ερωτήσεις να κάνετε για σύντομες απαντήσεις. Παρακαλώ κύριος Βίγκλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και εσάς. Καλή χρονιά και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία και εσείς ε, με τους συνεργάτες σας και με τη δική μας την Επιτροπή. Αυτό ποθούμε. Για τον αερόμπι, δύο παρατηρήσεις και ίσως και μία απορία. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαίος Επίτροπος να διαπραγματεύεται εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιζητήσει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ τη προώθηση κάποιων ζητημάτων που βρίσκονται στην αναπτυξιακή ατζέντα ή το πακέτο τη Ντόχα. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι να βρούμε έναν τρόπο και τα συγκεκριμένα επίπεδα όπου πρέπει να συζητηθούν και να τεθούν κάποια νέα ζητήματα. Εάν δεν συζητήσουμε αυτά τα νέα ζητήματα, θα χάσουμε ευκαιρίε. Θα χάσουμε ευκαιρίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, νομίζω ότι εάν στο Ναϊρόμπι υπήρχε ένα σαφές μήνυμα ότι ο ΠΟΕ είναι, στέκεται καλά στα πόδια του και μπορεί να δώσει αποτελέσματα, τότε πέραν πάσης αμφιβολίας, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσουμε και όπου μπορούμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπαθίες μας, τις διμερείς επαφές. Οι δύο αυτές διαδικασίες δεν είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Υπάρχουν σημαντικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και στο πρόγραμμα εργασίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ερχόμενο διάστημα επίσης υπάρχουν επιχειρήματα για να ξεκινήσουν νέες διμερείς διαπραγματεύσεις. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Βλέπετε κάποια αντίφαση ή ακούσατε στις συζητήσεις σας στον Ταβός ή μετά τον Αιρόμπι. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα βεβαίως και ήταν και γιορτές, ε, διακοπές. Αλλά οι δράσεις ε, για την φάση μετά τον Αιρόμπι είναι ανταγωνιστικές ε, και αντίθετες ως προς τις διμερείς συμφωνίες και τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιφάσκουν και για την αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική παρουσία αυτή. Και όταν μιλάμε και για την κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, καλό θα ήταν από την πλευρά της Επιτροπής να μιλήσει και να επιρρώσει αυτή την κοινοβουλευτική διάσταση που θα μπορούσε να είναι και μία από τις οδούς που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ε, ευχηθώ καλή χρονιά στην ε, Επίτροπο και να τη συγχαρώ για την εντατική και τόσο σκληρή δουλειά που έκανε κατά τη διάρκεια της υπουργικής διάσκεψης και είχα την ευκαιρία να το ε, διαπιστώσω αυτό η Μία από τις επιτυχίες είναι αυτό που ακούσαμε για την κατάργηση των εξαγωγικών γεωργικών επιδοτήσεων. Αλλά στη συμφωνία νομίζω δεν έχει δοθεί ειδικό βάρος ε, όσο θα έπρεπε στις τεχνολογίες προφορίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εμείς δεν καταφέραμε να το μεταλαμπαδεύσουμε, να καταλάβουμε τι ε, σημαίνει και πώς μπορεί αυτό να είναι υπέρ των καταναλωτών και των πολιτών εν γέννη. Τι θα γίνει τώρα μετά τον Ναϊρόμπι ποιοι θα είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι άξονες προτεραιότητες και το πρόγραμμα, το θεματολόγιο μετά τον Ναϊρόμπι. Όλες αυτές οι συμφωνίες που είναι ε, πολυμερούς χαρακτήρα, πώς θα συντονιστούν για να προχωρήσουμε υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ των ε, ισορροπιών που είναι πάρα πολύ εύθραυστες και το αναγνωρίζω. Θα ήταν τρομερό να μην υπάρχει συμφωνία, έτσι κι αλλιώς, αυτό θα ήταν όλεθρος και καταστροφή και δεν το συζητώ καθόλου, ε, αλλά ε, ε, νομίζω ότι η πρόοδος δεν ήταν και τεράστια στην ατζέντα της ανάπτυξης, ούτε για τα νέα στοιχεία που πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε. Τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα της ψηφιακής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πού πήγε αυτό και είναι κλειδί, διότι είναι παρόν στη ζωή μας, έχει έρθει για να μείνει και για να αναπτυχθεί και θα το έχουμε μπροστά μας. Άρα, χρειάζονται κανόνες για να τους εσπίσουμε εμείς. Πώς γίνεται αυτό, μπορούμε κάπως να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και πάλι σε πολυμερείς συμφωνίες ε, αναφέρομαι. Ευχαριστώ. Διαμά. Um, ευχαριστώ, Επίτροπε. Ήμουν και εγώ στο Ναϊρόμπι και σας είδα τώρα που δουλεύετε. Ευχαριστώ για τις μεγάλες σας προσπάθειες. Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι συνθήκαμε στην Αφρική Χάθηκαν και πολλέ ευκαιρίε. Αν και πήγαμε καλά στην πληροφορική, 10% του παγκοσμίου εμπορίου είναι καλό για του καταναλωτέ. Αν και δεν ξέρω πόσο αυτό βοηθάει τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Μετά είχαμε το καθόδε ε, θέμα τη γεωργία. Πώ θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει να πω πάντω, επειδή ήμουν στο Νερόμπι και ήσασταν και εσεί, ε, κύριε Επίτροπε, πού βρίσκεται το πρόβλημα. Όταν έρχεται η ώρα να διαπραγματευτούμε σε πολυμερές επίπεδο, δεν το πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε τον ΠΟΕ, δεν πιστεύουμε το πολυμερές πλαίσιο. Βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες, πλησιάζουμε στο τέρμα και, και δεν φτάνουμε στη, στη, στην πηγή. Σαν να λείπει δηλαδή η τελική προσπάθεια να πετύχουμε κάτι στο πολυμερές εμπόριο. Έχω τρεις ακόμα τάκουλα. Σόλτς και ένας ακόμα Επίτροπε, Πρόεδρε, συνάδελφοι, ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για άλλη μια φορά που βρήκε χρόνο να ενημερώσω την Επιτροπή μα σήμερα για τα αποτελέσματα τη υπουργική Διάσκεψη στο Ναρέομπι το Δεκέμβριο πέρσι. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχει συμφωνία για την αναπτυξιακή ατζέντα τη Ντόχας. Αυτό το αποτέλεσμα δεν το περιμέναμε καθόλου με βεβαιότητα πριν ξεκινήσει η αντιπροσωπεία για τον Ερόμπι. Δεν υπήρχε το κανένα τοποθέτησης τοποθέτηση όταν προσγειωνόμασταν στην Αφρική. Είναι ζωτική σημασία για το διεθνές εμπόριο, ιδίω όταν μιλάμε για μεγάλες οικονομίες της αγοράς και ευρωπαϊκές χώρες. Η χρήση του να πάυσουν οι επιδοτήσει λόγου χάρη ήταν σίγουρα ένα βήμα θετικό, ένα βήμα προόδου. Ε, Όμως ε, έτσι θα μπορέσουν πραγματικά να λειτουργήσουν εύρυθμα οι αγορές. Δεν θέλω βέβαια να μειώσω το νόημα των διαπραγματεύσεων που έγιναν επί 14 χρόνια στα πλαίσια του γύρου της Δόχας, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντοτε κατά των επιδοτήσεων. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στο Ναϊρόμπι μας δείχνει ότι οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν πραγματικά να διαπραγματευτούν και να υποχωρήσουν και ενδεχομένως σε ένα βαθμό να επαναχωρήσουν σε σχέση με τις ε, προηγούμενες θέσεις τους. Αυτό το μήνυμα πρέπει να δώσουμε προς τους πολίτες μας, έχοντας υπόψη τι ανταποκρίσεις και απαντήσεις είχαμε στις προηγούμενες φάσεις και το τι έχει γίνει και στις διαπραγματεύσεις της Διατλαντικής Συμφωνίας. Ε, μια άλλη πτυχή που δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για την συμφωνία περί των επιδοτήσεων από την ευρωπαϊκή και όλα οπτική γωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο εταίρος εκείνος που πρέπει να κάνει τις μεγαλύτερες αλλαγέ για να εφαρμόσει τη νέα συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρησιμοποιήσει εξαγωγικέ επιδοτήσεις εδώ και κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα σε πρακτικότερο επίπεδο. Το να οργανωθεί η υπουργική διάσκεψη στην Αφρική ήταν ένα σαφέ μήνυμα ότι όλα τα μέλη του ΠΟΕ ε, υποστηρίζουν την ίση συμμετοχή των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών στην οικονομία τη αγορά. Το να διοργανωθεί μια τέτοια υπουργική διάσκεψη και γενικότερο η διοργάνωση τέτοιων είναι πολύ σημαντικό. Ε, δεν είναι απλό ούτε καν το πρακτικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Πρέπει παρόλα αυτά να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι στο Ναϊρόμπι. Οι ενημερώσει τη Επιτροπή ήταν δύσκολο να διοργανηθούν, καθώ οι εκπρόσωποι τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου ε, βρίσκονταν σε διαφορετικά ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία ήταν μακριά μεταξύ τους και η πρόσβαση των μεν στα ξενοδοχεία των δε ήταν ε, περιορισμένη και ελεγχόμενη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικά μέσα για τέτοιου είδου συζητήσει. Η δική μου λοιπόν πρόταση είναι να λάβουμε υπόψη τι συνδικέ αυτέ συνθήκε και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε γενικά την κατάσταση. Θα ήθελα να πω το εξή. Όταν γίνονται οι προπαρασκευαστικέ, όταν θα γίνουν οι προπαρασκευαστικέ για την επόμενη υπουργική διάσκεψη, αυτό το σημαντικό στοιχείο να ληφθεί υπόψη, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να ενημερώσει καλύτερα του ευρωβουλευτέ. Αυτή ήταν η πρώτη μου, η πρώτη μου συμμετοχή σε υπουργική διάσκεψη και για μένα συνολικά ήταν μια εμπειρία πολύ θετική. Κυρίω λόγω του θετικού τη αποτελέσματο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Χέλμουτ Σόλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Μάσον που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να μας δώσετε τη δική σας ανάλυση του αποτελέσματος της Υπουργικής Διάσκεψης και της Έκφασης. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Συζητούμε αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούμε εντόνως όλους τους υπεύθυνους πολιτικούς να κάνουν κάτι, ό,τι μπορούν για να εκριζωθούν οι αιτίε που οθούν τους ανθρώπους ε, να ε, φεύγουν από τις πατρίδες τους. Ένα σύντομο σχόλιο για το προσφυγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον καιρό. Όσο συζητούμε λοιπόν ε, το αποτέλεσμα της υπουργικής διάσκεψης ε, του ΠΟΕ θα πρέπει να ζήσουμε και αυτή την πρόκληση. Πώς θα ε, αναδομήσουμε τις διεθνείς πολιτικές, το διεθνούς εμπορίου, θα το συνδέσουμε με αναπτυξιακές πολιτικές, πολιτικές εξωτερικής πολιτικής για να δούμε τι γίνεται στις χώρες που μαστίζονται από φτώχεια και ο κόσμος δεν έχει άλλες επιλογές παρά να φύγει από τη χώρα του. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο κατά την άποψή μου. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι βεβαίως υπήρξε ένα αποτέλεσμα στην υπουργική διάσκεψη, αλλά είναι κάπως ένα ανεφέλωμα αυτό. Πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και μπρος πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις του γύρου ανάπτυξης της Ντόχα. Θα δώσουμε την ευκαιρία στις χώρες αυτές να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο, σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα. Θα ανοίξουμε νέα ζητήματα που βεβαίως είναι επιτάπητος. Καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν είναι δεσμευτικά όλα αυτά για τις χώρες, δεν έχουν σαφείς υποχρεώσεις, θέλω να ρωτήσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκέφτεται να συνεισφέρει για να λυθεί αυτή η προφανής ε, αντίφαση. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά συμφωνώ με όλους εκείνους τους συναδέλφους που λέγουν ότι βεβαίως χρειαζόμαστε κάποια ε, κοινοβουλευτική διάσταση και στον ΠΟΕ. Και κάποιος μου είπε ε, βέντω στο, στο ε, Ναϊρόμπι ότι συμφωνεί να υπάρξει και ένας οδικός χάρτης για το πώς μπορεί κανείς να προχωρήσει σε αυτό. Ο κύριος Μπούχνερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Έχω μερικές ερωτήσεις. Ο καιρός ε, του ε, γύρου της Δόχας, το πρακτικό ρόλο το δικό σας έχει παρέλθει ουσιαστικά. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει τι μέλη γενέστε στην κατεύθυνση αυτή, ποιο είναι το επόμενο βήμα και σχετικό με το προηγούμενο. Δεν ήταν όλοι πανευτυχεί από το αποτέλεσμα τη Υπουργική διάσκεψης, ιδιαίτερα κάποιες αναπτυσσόμενες χώρε και χώρε από τις πιο φτωχέ του κόσμου, οι κυβερνήσει του σε πάση περιπτώσει. Και σε σχέση με αυτό και κάποιες ΜΚΟ. Εσεί δεν διαβλέπετε εκεί κανένα κίνδυνο. Δηλαδή να κινόμαστε τελείως ερήμην ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού και να κάνουμε μια πολιτική υπέρ των πλουσίων χωρών, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τις φτωχότερε. Η κυρία ε, Μπικέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την Επίτροπο που ήρθε να μας ενημερώσει και για τα όσα έκανε κατά την Υπουργική Διάσκεψη στο Νερόμπι. Συνολικά, νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα μετριοπαθές παρά την αρχικά άκαμπτη στάση των ΗΠΑ. Για την Ντόχα τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Παρόλο που στο τελικό κείμενο δεν υπήρχε μνήα του γεγονότος πριν αποφύγουμε τις, τον πολλαπλασιασμό των διμερών και περιφερειακών ε, συμφωνιών, κάτι που θα σημαίνει ότι το σύστημα του ΠΟΕ γίνεται λίγο ένα σύστημα à carte Όμω υπάρχουν κάποια σημεία που είχαν συζητηθεί ήδη πριν από τον Ναϊρόμπι και ακόμη παρέμενουν εκκρεμοί. Όπως ορισμό των αναπτυσσόμενων χωρών. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία δεν μπορούν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Και η ερώτησή μου προς εσάς, δεδομένης και της επικαιρότητα είναι πώς βλέπετε το μέλλον. Και ολοκληρώνω, επειδή χρόνος δεν υπάρχει. Thanks a Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, βλέπετε και από τον κύριο Τάκουλα ε, ακούσατε πώς έχει βελτιωθεί η ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα στην τελική φάση μιας διαπραγμάτευσης και πραγματικά πρέπει να πω ότι υπήρξε κάποια συζήτηση ακόμα και μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ότι χωράει βελτίωση αυτή η επικοινωνία μέσα Φεβρουαρίου θα συναντήσουμε κυρία Πίτροπε τους ομολόγους μας από άλλα κοινοβούλια των κρατών μελών ε, του ΠΟΕ. Τι θα μας συμβουλεύατε να συζητήσουμε σε αυτό το γύρο του Φεβρουαρίου. Thank you, Thank Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, θα είμαι σύντομη ως προς τον κύριο Βίνκλα και το ερώτημά του. Ε, ναι, επέστρεψε από το Νταβός. Είναι ένα κλειστό φόρουμ όπου συνάζουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλη επιρροή. Οι επιχειρηματίε που ήταν εκεί, αλλά και η ΜΚΟ, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που ήταν εκεί, που δεν είναι εκπρόσωποι τους πάντες φυσικά, ήταν λελογισμένα αισιόδοξοι. Και είπαν ότι ο ΠΟΕ έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν πετύχαμε τα πάντα, ήταν καλή συμφωνία που αποδεικνύει μας πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΟΕ ζει. Κατά τα άλλα, στις παγκόσμιες αγορές σοβεί αβεβαιότητα. Άλλωστε αυτά τα οποία συζητήσαμε, Γεωργία για παράδειγμα, είναι μέρος και μόνο της παγκόσμιας ατζέντα. Συνεπώς, οι περισσότεροι, πολλοί τουλάχιστον, παίκτες στο διεθνές επίπεδο θέλουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Θα προχωρήσουμε πολυμερώς και διμερώς. Το θέμα είναι βεβαίως όλα να συνάδουν με το υφιστάμενο πλαίσιο του ΠΟΕ. Θα μας βοηθήσει αυτό και θα αναπτύξουμε και νέα πρότυπα, τα οποία θα φέρουμε πιο κοντά για να γίνουν τμήματα του πολυμερούς πλέον πλαισίου. Το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Τώρα η κοινοβουλευτική διάσταση που ανέφερε και ο Στάκουλα και ο Πρόεδρος φυσικά είναι πολύ σημαντική. Σήμερα δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεκαθαρίσει τι σημαίνει αυτό στην πράξη, αλλά σίγουρο είναι να συζητήσουμε και να είστε και εσείς σε αυτή τη συζήτηση. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ίσως να χρειαστούμε μια πιο άτυπη συζήτηση. Ο τρόπος πάντως με τον οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση στον Ναϊρόμπι και να σας πω, να σας εξομολογηθώ ότι ε, νόμιζα ότι θα τελειώσουμε σε 20 λεπτά και βγήκαμε έξω μετά από 26 ώρες. Ήταν εκεί η Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κίνα, η Ινδία και φυσικά εκπρόσωποι των Αφρικανικών κρατών, κυρία Μοχάμερ βεβαίω ε, από τις Αφρικανικές χώρες. Ε, και να σου πω την αλήθεια, δεν υπήρχε χρόνος για ενημέρωση. Το Συμβούλιο ήταν καλύτερα πληροφορημένο από εμά. Αλλά όπω είπε και εσύ κύριε Τάκουλα, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχαν έγγραφα, δεν ήταν καλή η προετοιμασία. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την διαδικασία πολύ νωρίτερα από την επόμενη σύνοδο το 2017. Θα βελτιωθούμε. Ούτε μάλιστα το Συμβουλίο πρέπει να σας πω ήταν ευχαριστημένο από... με την έλλειψη επαφών. Έχασαν δύο ολοκληρές μέρες εκεί. Λοιπόν, πώς θα ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση. Αυτό είναι ένα πράγμα. Τώρα, αφού γραζόμαστε απλώς, να δούμε τι θέματα πρέπει, μπορούμε και πρέπει να προσθέσουμε στην ατζέντα. Είναι λίγο νωρί. Δύο εβδομάδες μετά να αρχίσουμε να λέμε να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Όχι. Είπατε για το ψηφιακό εμπόριο ή το ηλεκτρονικό εμπόριο. Βεβαίω, Είναι ο προφανή υποψήφιο, το προφανέ επόμενο βήμα. Άλλοι μιλούν για τι επενδύσει. το τοπικό, περιφερειακό περιεχόμενο κλπ. Όλα αυτά ισχύουν. Όμως ας κοντοσταθούμε, ας αφουγκραστούμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη συμφωνία και ας κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη γιατί δεν θα ορμήξουν όλοι να συμφωνήσουμε ό,τι και αν φέρουμε στον ΠΟΕ. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε συζητώντα σιγά σιγά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, για παράδειγμα, είναι ένα ε, ελέφαντα. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημά του μία νυχτή. Α δούμε λοιπόν τι έχουμε στο τραπέζι. Α δούμε τι θα συζητήσει το Συμβουλίο την επόμενη εβδομάδα και θα έχετε κι εσεί τι δικέ σα ιδέε γιατί η κοινοβουλευτική διάσταση και η συζήτηση είναι πολύ σημαντική βεβαίω. Κύριε Μακλάφεν, για την Γεωργία συμφωνώ. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει έχουμε πετύχει περισσότερα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αν δεν είχαμε πάει επί τόπου, δεν είχαμε πετύχει συμφωνία. Διότι οι χώρες με τους μεγαλύτερους ε, δισταγμούς, ε, αν δεν ήταν εκεί δεν είχαμε συμφωνήσει ποτέ. Αν είχαμε μείνει εδώ ή στην Γενέβη, αν η ζήτηση αυτή είχε γίνει αλλού, δεν είχαμε προχωρήσει σε καμία περίπτωση. Προχωρήσαμε με την ατζέντα της Δόχα. εκκρεμούν φυσικά ζητήματα που άπτονται της γεωργίας, υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τη συμμετοχή του δημοσίου, του public stockholding. Ε, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει τόσο σκεπτικισμός όσον αφορά τον πολυμερή χαρακτήρα αυτών των συμφωνιών, περισσότερο εδώ τουλάχιστον σε σχέση με άλλους. Ε, Πάνω 164 χώρες δεν συμφωνούν εύκολα, ούτε προχωρούν εύκολα προς την διακατεύθυνση. Αλλά αυτό είναι και το πλεονέκτημα του ΠΟΕ. Προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε μια ισορροπία, να φέρουμε όλους τους διστάζοντες μαζί μας. Ξεκινούμε κάθε φορά να δουλεύουμε λίγοι, πολύ λίγοι και προσπαθούμε ότι πετυχαίνουμε να το φέρουμε πιο κοντά στο πολυμερές πλαίσιο, να αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα. Και σωστά συμφωνώ, το εμπόριο διδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα, όμως αν το συνδυάσουμε με άλλες έξυπνες πολιτικές ανάπτυξης, με πολιτική συνεργασία και με εμπόριο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα έχουν πλέον οικονομικούς τουλάχιστον λόγους να μεταναστεύσουν. Και το τόνισε αυτό στη στρατηγική εμπορία για όλους. Ότι τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες στο Ναϊρόμπι και αυτέ δεν ήταν ευχαριστημένε, αλλά αυτά τα οποία συμφωνήσαμε για την Γεωργία ήταν καλά για πολλέ αφρικανικέ χώρε. Για τον Μπαμπάκι πετύχαμε μια συμφωνία η οποία δίνει πρόσβαση στι διεθνεί αγορέ για χώρε που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το βαμβάκι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι πήγαμε να συζητήσουμε μόνο θέματα που συμφέρουν ή ενδιαφέρουν του Ευρωπαϊού και του Αμερικανού. Και έπαιγε το τι είναι αναπτυσσόμενη χώρα ε, δεν θα πρέπει να επισκιάσει την ουσία της συζήτησης γιατί κάποιες χώρες αυτοπροσδιορίζονται ως αναπτυσσόμενες. Ξέρουμε τα κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις LDC. Οι άλλες είναι αναπτυσσόμενες χώρες και φυσικά λένε ότι καμιά φορά πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση που έχουν οι LDC, οι πολύ φτωχέ χώρες. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι Άλλο να έχει κάποιο πρόβλημα ανάπτυξης και να είσαι μια ισχυρή οικονομικά χώρα και άλλο να είσαι μια από τις πολύ φτωχέ χώρες. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι είμαι φτωχός όταν είσαι κάπου στη μέση. Γι' αυτό δεν υπάρχει λύση. Όμως αποδείχθηκε ένα από τα πλέον ακαθόδη προβλήματα. Χάρη στην πολιτική συνεργασία πάντω θα προχωρήσουμε. Ε, έχετε πάντως επαναλαμβάνω δίκαιο που το εντοπίζετε αυτό ως ένα από τα βασικά προβλήματα. Δεν έχουμε βρει τρόπο ακόμη, δεν έχουμε βρει λύση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Α, για το χρονοδιάγραμμα λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνήθηκε τι θα κάνουμε ας πούμε σε 6 μήνες από τώρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον και είναι ρεαλιστικό αυτό, 6 μήνες. Είμαστε έτοιμοι να, να ζητήσουμε από τους πρέσβεις στη Γενέβη να ορίσουν την ατζέντα για το μέλλον. Δεν συμφωνήσαμε για ημερομηνίε, λέει η κυρία Μάλστρομ. ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα από σήμερα, από την επαύριο των συνομιλιών, για την υλοποίηση, να καταργήσουμε τι εξαγωγικέ επιδοτήσει, το οποίο θα είναι καλό για εμά, για τον Καναδά, για την Ελβετία. Προετοιμάζουν και εκεί τι κοινοβουλευτικέ του ε, διαδικασίε. Είπαμε ότι οι πρέσβει, οι την πρόσωπη στην ε, Γενέβη θα συνεχίσουν να εργάζονται από των θεμάτων, αλλά χρειάζονται πολιτική καθοδήγηση. Διότι υποτίθεται ότι το παλεύουμε εδώ και χρόνια, πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η κυρία Ζεβέδο είπε ότι κρατημέλη και ο ΠΟΕ Πρέπει να καθίσουν γύρω το τραπέζι, να συζητήσουν νέε ιδέες, να δούμε πώς μπορούμε να προσετεριστούμε ε, και τις υπόλοιπε χώρε πέρα από αυτές που πρωτοπορούν. Τον Ιούνιο στο Παρίσι έχω μια συνάντηση στον Νόσα. Πολλέ από τι χώρες αυτές θα είναι εκεί και θα τα πούμε και στο περιθώριο της ε, διάσκεψης και έχουμε και το G20 για το εμπόριο στην Σανγκάη μέσα Ιουλίου όπου θα συζητήσουμε και πάλι τα ίδια θέματα και την επόμενη εβδομάδα βεβαίω στο άτυπο συμβούλιο. Το θέμα είναι στη σε διάταξη μαζί με τον Αζεβέδο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε τα θέματα χωρίς να υπάρχει όμως καμία συγκεκριμένη προθεσμία. Ευχαριστούμε πολύ Επιτροπέ πολύ καλό το υλικό που μας δώσατε για να συλλογιστούμε το πώς θα διαμορφωθεί η διαδικασία στη φάση μετά τον Ναϊρόμπι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Παρουσίαση από την ε, Ολλανδική Προεδρία, την Υπουργό Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και να καλωσορίσω την κυρία Πλούμεν, ακριβώς, Υπουργό Εξωτερικού μπορεί και δείξει και Συνεργασίας της Ολλανδίας και προφανώς καλύπτει και τα θέματα ανάπτυξης στο Υπουργείο σε αυτά που ενδιαφέρουν εμάς. Η Προεδρία έχει ξεκινήσει και πριν από την Προεδρία για το πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει αξία, υπεραξία και ε, είναι πολύ καλό βήμα αυτό ε, για ένα σύστημα εμπορίου του 21ου αιώνα σε συνθήκες δικαιοσύνης. Έτσι το βλέπω εγώ και ελπίζω από κοινού να ε, διαβούμε το δρόμο αυτό το επόμενο εξάμεινο και να το συνεχίσουμε. Έχουμε μια νομοθεσία που μας απασχολεί, η νομοθεσία κατά των βασανιστήριων ή τα ε, θέματα των ε, μεταλλευμάτων από εμπόλεμες ε, ζώνες και κάποιες συμφωνίες που μας συνοδεύουν, είτε αυτή είναι TTIP, είτε συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά ή συμφωνίες εταιρικής σχέσης με αφρικανικές χώρες. Και βεβαίως και το θέμα της Ουκρανίας αλίμονο και των ε, σχέσεων της Ανατολικής Γειτονίας και θέματα μετανάστευσης επίσης και αυτό που μόλις συζητήσαμε τι συνέχεια θα δοθεί στον ΠΟΕ. Όλα αυτά τα ζητήματα θα κυριαρχήσουν ε, το επόμενο διάστημα την Άνοιξη. Κυρία Υπουργέ. Η κυρία Πλάουμεν θα κάνει ε, μια εισαγωγή και μετά θα πάρουν το λόγο πολιτικές ομάδες. Οχτώ ήδη έχουμε και αν θέλουν και άλλοι οι βουλευτές να μιλήσουν, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να είναι σύντομες για να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Τρία τέταρτα χρόνο έχουμε. Υπουργέ, έχετε το λόγο κυρία Πλάουμεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι στα γαλλικά Υπουργό και στα αγγλικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ενώπιον σας εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι όταν ένας υπουργό μιας εθνικής κυβέρνησης ε, έρχεται ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να έχουμε επαφές με ευρωβουλευτές. Σας είπα ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που έχω να συζητήσω θέματα ε, που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Διότι το εμπόριο δεν έχει να κάνει μόνο με τις κόκκινες γραμμές ή με τους δασμούς. Το εμπόριο έχει να κάνει και με τις θέσεις εργασίας και με τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, για καινοτομία. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς εμείς οι Ευρωπαίοι ε, συνδεόμαστε και συνεργαζόμαστε με άλλες ε, εμπορικές οντότητες, με λαούς και με χώρες σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, τι εννοώ αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε μόνο το δικό μας δυναμικό, αλλά να συνεργαζόμαστε με άλλους έτσι ώστε από κοινού να βελτιώνουμε τον κόσμο. Και όπως ε, ήδη είπε ο πρόεδρος ο κ. Λάγκεν, δεν είμαι μόνο υπουργό εμπορίου, αλλά είμαι και υπουργό αναπτυξιακής βοήθειας. Και τώρα που ε, συνδέονται τα πράγματα. Μια μητέρα στο Παγκλαντές που ε, ράβει ένα μπλουζάκι και μια μητέρα στο Άμστερνταμ που ζω εγώ το αγοράζει για το παιδί της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την πολυδιάστατη και πολύπλευρή προσέγγιση. Αναλάβαμε την Προεδρία οι κάτω χώρε σε καιρού, θα έλεγα, πραγματικά ε, δύσκολου με προκλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό, Ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να συνεργαζόμαστε ω Ένωση, ω Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε τον εξτρεμισμό, ε, ανίποτη και πρωτοφανή αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Η κατάσταση είναι περίπλοκη και εύθραυστη σε πολλά από τα σύνορά μας. Σε αυτούς λοιπόν τους χαλεπούς καιρούς θα έλεγα και θα πρότεινα ε, να έχουμε στο πλευρό μας παραστάτη και τέρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορεί η Ευρώπη να ε, έχει αποτελέσματα για τους πολίτες ε, πάντα σεβόμενοι τις αρχές και τις αξίες. Εμείς θα είμαστε μία δραστήρια προεδρία. Δεν νομίζω να περιμένετε τίποτα διαφορετικό από εμάς, αλλά θα είμαστε και ρεαλιστές. Γι' αυτό διακρινόμαστε εμεί οι Ολλανδοί και μα γνωρίζει ο κόσμο. Θέλουμε χειροπιαστά αποτελέσματα το επόμενο εξάμεινο σε όλου του ομίλου που σα ανέφερα και τα θέματα που θα μα απασχολήσουν σήμερα εδώ, ειδικότερα του εμπορίου. Η Προεδρία μας θα εργαστεί για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να εστιάζει στα βασικά, στα θεμελιώδη, να συνδέεται γενικά με την κοινωνία και ε, να κάνει τους λαούς να συμμετέχουν και τους πολίτες με τρόπο ενεργό. Βεβαίως μιλώ εδώ και για ΜΚΟ και για εταιρείες και πάντα σεβόμενοι την αρχή της διαφάνειας. Και παρακαλώ το επόμενο διάστημα, το επόμενο εξάμεινο να μας ε, ε, εγκαλείτε και είμαστε υπόλογοι σε αυτό. Η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει και αυτή είναι ευχάριστη είδηση και καλό ε, είναι από κοινού να συνεργαστούμε για να διατηρηθεί αυτή η θετική τάση έτσι ώστε η οικονομική ε, ανάπτυξη, η μεγέθυνση να γίνεται χωρίς αποκλεισμούς, να υποφελούνται οι πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ανάπτυξη να δημιουργεί θέσεις εργασίας για όσο γίνεται περισσότερους πολίτες. Και βεβαίως ε, θέλουμε να προωθήσουμε και την καινοτομία από μια υφόρο ανάπτυξη. Να ενθαρρύνουμε τους πάντες να συμμετέχουν σε αυτή την ακριβώς συμμετοχική οικονομία, μικρομεσαίες επιχειρηματίες αλλά και μεγαλύτεροι όμιλοι, εταιρείες, πολίτες και χρειαζόμαστε στο πλευρό μας την κοινωνία των πολιτών, να αναλάβει και το δικό της ρόλο. Τώρα, εγώ δεν χρειάζεται να σας πείσω εσάς, τα γνωρίζετε εδώ σε αυτή την ομίγυρη. Η υπόθεση του διεθνούς εμπορίου είναι βασικό συστατικό και παράγον αυτής της οικονομικής ανάπτυξης που θα είναι και διαρκής και χωρίς αποκλεισμούς. Και αυτές είναι και προτεραιότητές μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να τις συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Τις προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας. Τέσσερις είναι αυτές για το εμπόριο. Πρώτο είναι η ε, ε, ε, τόνωση της ένταξης της ολοκλήρωσης μάλλον της πολιτικής εμπορίου και της πολιτικής αναπτυξιακής βοήθειας για να προωθηθεί εφορία. Ο κύριος Λάγκελ αναφέρθηκε σε μια διάσκεψη του Δεκεμβρίου και θα επανέλθω στη συνέχεια. Δεύτερη προτεραιότητα, να προχωρήσει η συζήτηση για τη μετά το Ναϊρόμπι εποχή και από ό,τι κατάλαβα μόλις το συζητούσατε με την Επίτροπο την κυρία Μάλμστρομ που διαπραγματεύτηκε εξ ονόματός μας τη συμφωνία αυτή η συζήτηση για την εποχή μετά τον Αιρόμπι έχει και την εξή σημασία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την υλοποίηση των όσων αποφασίστηκαν στον Παλί και τον Αιρόμπι, αλλά έχει να κάνει και με το μελλοντικό ρόλο του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τρίτη προτεραιότητα είναι να διευκολυθούν ε, οι ε, συνεχιζόμενες διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με μια ειδική εστίαση και αυτό δεν θα σας εκπλήξει στο TTIP, ε, ΣΥΤΑ και τις συμφωνίες με την Ιαπωνία και κάποιες άλλες οικονομικές συμφωνίες με χώρες της Αφρικής. Το τέταρτο, χωρί αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό και ξέρω ότι πολλοί από εσά συμμετείχατε στην προώθηση αυτών των δύο νομοθετικών συζητήσεων, το ένα έχει να κάνει ε, με την καταπολέμηση των ε, βασανιστήριων και των άλλων με τα μεταλλεύματα από τις εμπόλεμες περιοχές. Να σας πω δύο λόγια, όχι πάρα πολλά, γιατί πραγματικά περιμένω να ακούσω ε, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Οι βιώσιμες παγκόσμιες αλυσίδες αξιών είναι πάρα πολύ σημαντικές για μια αηφόρο οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση παγκοσμίω. Τι εννοώ, Υπάρχουν πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός της Ένωσης ε, που συνδέονται με αυτές τις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και τη δυνατότητα και το δυναμικό και τα εργαλεία και, και τους μοχλούς. Ε, είμαστε η μεγαλύτερη αγορά, 500 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουμε κάποια διαπραγματευτική δύναμη, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και αυτό άμεσα επηρεάζει ανθρώπους που ζουν στην άλλη άκρη του πλανήτη. Στις 7 Δεκεμβρίου είχαμε μια διάσκεψη για το θέμα αυτό, αλλά για να το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, εγώ θα διοργανώσω ε, μια άτυπη ε, σύνοδο Υπουργών Εμπορίου και ε, Αναπτυξικής Βοήθειας στις 2 Φεβρουαρίου. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό, κοινή υπουργική συνεδρίαση και ελπίζω να δοθεί και συνέχεια. Γιατί αν δείτε τα νομοθετικά ζητήματα που μας περιμένουν τους επόμενους έξι μήνες και για τα βασανιστήρια και για τα μέταλλα από τις εμπόλεμες περιοχές ε, θα καταλάβετε ότι ε, ε, σχετίζονται και με το εμπόριο και με την αναπτυξιακή βοήθεια και τα υπόλοιπα που σας έλεγα. Η έκβαση λοιπόν αυτών των διασκέψεων θα μας βοηθήσει να στρώσουμε μια στρατηγική για ε, την ε, παγκόσμια ανάπτυξη και με την εξωτερική διάσταση με ένα πρόγραμμα δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ένα κώδικα δεοντολογίας για τους επιχειρηματίες με υπευθυνότητα. Στον Ταβός, ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα κυριάρχησε αυτό το θέμα. Χρειάστηκε να το καταλάβει αυτό ο επιχειρηματικό ε, κόσμος και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζω να κάνει βήματα. Η δεύτερη προτεραιότητα μετά τον Αερόμπι, ε, μάλλον δεύτερη προτεραιότητα είναι ο ΠΟΕ μετά τον Αιρόμπι. Οι ε, κάτω χώρες πάντα ήταν πάρα πολύ ενεργό μέλος στον ΠΟΕ, ανέκαθεν, Διαπραγματευόμαστε βέβαια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντα και θα συνεχίσουμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο. Καλωσορίζουμε την ΚΑΝΠΗ συμφωνία που επετεύχθη στη 10η Υπουργική Διάσκεψη το Δεκέμβριο στο Ναϊρόμπι. Κατά την άποψή μου η κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων στη Γεωργία είναι από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του Νερόμπι και θα είναι προς όφελος όλων των μέλων του ΠΟΕ με κύρια έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες. Βλέπω εδώ τις ομάδες που είναι παρούσες και ξέρω και κατανοώ ότι πολλοί από εσά πιέσατε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, άλλο χαρακτηριστικό της συμφωνίας ήταν η Συμφωνία ΙΤΑ για, για προϊόντα ε, ε νέων τεχνολογιών ε, Πληροφορική μέχρι και 20 προϊόντα, 200 ε, συγγνώμη. Δεν ήταν εύκολο να συμφωνηθεί αυτό και έχει να κάνει με την περίοδο και τη συζήτηση που θα γίνει για την εποχή μετά τον Ναϊρόμπι. Προσκάλεσα τους συναδέλφους ε, στο Συμβούλιο να το συζητήσουμε αυτό μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 2 Φεβρουαρίου σε ένα δείπνο. Εκπρόσωποι του ΠΟΕ θα είναι εκεί, ε, του ΟΑΣΕ, του, του ΟΣΑ συγγνώμη, και της ΟΥΝΚΤΑΤ είχαν την καλοσύνη να δεχθούν την πρόσκληση, θα έρθουν και θα παρουσιάσουν ε, τις απόψεις τους. Θέλω επίσης να ακούσω τις απόψεις σας γι' αυτό, προσβλέπω σε αυτό και ξέρω ότι είχατε μεγάλη συζήτηση με την Επίτροπο Μάλστρομ. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να έχετε και κάποια σχόλια για τη δική μας Προεδρία και ερωτήσεις. Για τις διμερείς τώρα διαπραγματεύσεις, τρίτη προτεραιότητα για την Προεδρία μας. Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στο TTIP ε, και τη διαπραγματεύση με την Ιαπωνία και ε, τη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι το TTIP. Η συμφωνία αυτή θα ωφελήσει τις οικονομίες μας μακροπρόθεσμα και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας, τις ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων αποσχόλησης και συνολικά την ευμάρειά μας. Στόχος μας και ακόμη είναι στόχος αυτός ε, να έχουμε μια σφαιρική εμπορική συμφωνία που να αφορά όχι μόνο τις προτιμησιακές δασμολογικές ρυθμίσεις αλλά και τους μη δασμολογικούς φραγμούς και επίσης να καθοριστούν κανόνες, πρότυπα ώστε οι δικές μας αξίες να εμφυσιθούν σε συμφωνίες που θα ωφελήσουν ευρύτερα την κοινότητα των εμπορευομένων και το μεγαλύτερο μέρος πολιτών που είναι δυνατόν παγκοσμίω. Έχουμε ήδη συζητήσει στο Κοινοβούλιο και άλλες προτεραιότητες και χαίρομαι που και εσείς συμμερίζεστε κάποιες από αυτές μαζί μας, ιδίως για την προστασία των επενδύσεων. Υπάρχει μια νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύστημα δικαστικό πρακτικής επίλυσης των διαφορών περί επενδύσεων. Οι ισχυρότερε θέσεις και φωνές που ακούστηκαν σε αυτό το κοινοβούλιο ήταν υπέρ αυτής της λύσης και όπως ξέρετε η Ολλανδική κυβέρνηση έχει στηρίξει την συγκεκριμένη επιλογή. Η συμφωνία TTIP δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τα πρότυπά μας για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την απασχόληση δεν θα είναι επιτυχής η έκβαση των διαπραγματεύσεων εάν αυτά τα πρότυπα και αυτές οι προδιαγραφές δεν γίνουν σεβαστά. Έχουμε εργαστεί και θα εργαστούμε σκληρά στο κεφάλαιο και στη διάσταση της διαφάνειας. Το Κοινοβούλιο γενικώ και η δική σας επιτροπή, η δική σας επιτροπή πιέζει ε, υπέρ αυτής της ε, προτεραιότητας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό η Προεδρία είναι μαζί σας. Για την Ιαπωνία. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις κοιτάζοντας όχι μόνο προς τα ε, αριστερά μας αλλά και προς τα δεξιά μας είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος, ο η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου η, Ιαπωνία και ελπίζω ότι οι διαπραγματεύσει θα ολοκληρωθούν φέτος μαζί τους. Η Προεδρία του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φανεί φιλόδεξη, αλλά και η Ιαπωνία θα πρέπει να φανεί πρόθυμη να κάνει μια πρόταση χειροπιαστή και εύκολη να υλοποιηθεί. Για τις οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης είμαστε υπέρ τέτοιου είδους κινήσεων και θα θέλαμε να υπογραφούν κάποιες από αυτές τις συμφωνίες, κάποιες από αυτές που ξεκίνησαν στην αρχή της χρονιάς, ιδίω με χώρες της Νοτιού και Ανατολικής Αφρικής. Θέλουμε να συνεργαστούμε με αυτές τις γεωγραφικές περιοχές και να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των συμφωνιών. Επίσης θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια οικονομικής συμφωνίας με χώρες της Δυτικής Αφρικής για την ε, διαφάνεια. Η διαφάνεια έχει να κάνει με τη διάθεση εγγράφων εδώ στους ευρωβουλευτές και σε βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το επίπεδο να απομυθοποιηθεί η διόλεκτος που χρησιμοποιείται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, διότι πολλές φορές εμείς ε, που βρισκόμαστε σε μια τέτοια αίθουσα καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας προς τη συγκεκριμένη ιδιόγλωσσα και αυτό κάνει και το Ολλανδικό Κοινοβούλιο λόγω χάρη. Θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να συζητάμε σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή και εύληπτη για τον καθένα που παρακολουθεί. Η Προεδρία λοιπόν θα κάνει μια σοβαρή και εντατικότατη προσπάθεια για να απλοποιήσει αυτή την ιδιόλεκτο και να χρησιμοποιεί εκφράσεις που όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν. Ελπίζω λοιπόν ότι θα σταθείτε στο πλευρό μου και τους ερχόμενους έξι μήνες θα βοηθήσετε να απομυθοποιήσουμε, να αποσαφηνίσουμε αυτή την εμπορική γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουν όλοι ποια είναι τα ωφέλη από το εμπόριο για τους ίδιους τους πολίτες. Τελευταία προτεραιότητα που ήθελα να αναφέρω, τα νομοθετικά ντοσιέ και ο κανονισμός κατά των βασανιστήριων. Ο πρώτος μας τριμερής διάλογος αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού ε, που διέπει την, ε, τις εμπορικές μας σχέσεις για ορισμένα αγαθά και που θα μπορούσαν να ε, χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν την θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές υποβάθμισης, ε, κακομεταχείρισης και απάνθρωπη συμπεριφορά. Θα συζητήσουμε ξανά με την, στην Προεδρία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο το θέμα αυτό και ήδη έχουμε συμφωνήσει για κάποιες βασικές προσθήκες όπως την ε, εκχώρηση αρμοδιοτητών και την τεχνική αρρωγή στα πλαίσια του οικονομισμού. Και βεβαίω εδώ η Προεδρία θεωρεί ότι έχει το καθήκον να καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν οι σωστέ συμβαστικέ λύσει. Αδειμονώ λοιπόν να συνεργαστούμε για να βρούμε αυτέ τι συμβαστικέ λύσει ακριβώ και έχω απόλυτη πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι ένα σημαντικότατο κανονισμό και σα ευχαριστώ για όλη σα τη δουλειά θα συνεργαστούμε. Δεύτερο νομοθετικό θέμα που μας απασχολεί είναι τα ορυκτά των συγκρούσεων. Εξίσου σημαντικό θα έλεγα γιατί επηρεάζει τόσους ε, πολλούς πληθυσμούς ανά την Ιφίλιο, κάποιους που δεν έχουν ε, δυνατότητα να υψώσουν τη φωνή τους όπως έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό, σε αυτό το κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο ως Προεδρία. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί όθηση για να ακουστεί η φωνή και αυτών των ε, ανθρώπων και να εκπροσωπηθούν στις συζητήσει μας. Ο τριμερής διάλογος δεν θα είναι εύκολος, αλλά υπάρχει προθυμία από όλες τις πλευρές, από το Συμβούλιο, από το Ευρωκοινοβούλιο, από όλους να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα και παρακαλώ βοηθήστε και εσείς την στενή μας αυτή συνεργασία για να έχουμε ένα αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Όχι γιατί εμείς είμαστε το ζητούμενο ως Ολλανδική Προεδρία, αλλά γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Και θέλουμε να λάβουμε αποφάσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ε, ASAP για να πάψει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, του πληθυσμού να υποφέρει. Τώρα, η το οικονομικό καθεστώς της Κίνας ως προς την αγορά, ένα άλλο σημαντικό θέμα επιτάπητος, ιδανικά το Συμβούλιο θα έπρεπε να υιοθετήσει μια θέση επί του θέματος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και ο τριμερής διάλογος να γίνει κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να καταθέσει μια πρόταση. Φαντάζομαι θα μας υποστηρίξετε και θα συμφωνήσετε, εμείς θα πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της αυτή. Ελπίζουμε ότι θα ετοιμάσουν και μια μελέτη αντικτύπου για να είμαστε πλήρως ενημεροί για το θέμα στις συζητήσεις μας. Ο στόχος είναι η διαδικασία να εκκληθεί ως το δυνατόν πιο ομαλά. Ε, ενίκη συμπεράσματο να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, αφοσίωση με την οποία εξετάζετε όλα τα ζητήματα τα οποία ανέφερα. Θα συνεργαστούμε και μάλιστα εντατικά. Θα είμαστε στη διάθεσή σας, στη διάθεση του Συμβουλίου, στη διάθεση των πολιτών. Ε, και όλων των ευρωπαϊκών κρατών βεβαίως ε, στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά το έργο της Προεδρίας. Εγώ ευχαριστώ Υπουργέ. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, οι πολιτικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και σχόλια. Οκτώ πολιτικές ομάδες έχουμε. And if we want to have... Εάν θέλετε να μιλήσουν και άλλοι βουλευτές, παρακαλώ να το έχετε αυτό υπόψη. Να είστε σύντομοι. Το, όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ο κύριος Γκασπάρη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που έχουμε σήμερα την ευκαιρία αυτή να ανταλλάξουμε απόψει μαζί σα. Εγώ έχω πολλέ επιφυλάξει όταν φέρνει πάρα πολλέ προτεραιότητε μία προεδρία. Και δυστυχώ, ε, και σήμερα αυτό ακούμε και το διαπιστώνω με ανησυχία, γιατί όταν έχει τόσε πολλέ προτεραιότητε, ε, δεν μπορεί να είναι τα πάντα προτεραιότητε, κάπου πρέπει να βάζει κέντρα βάρου. Αλλιώ υπάρχει ο κίνδυνο τα πράγματα να πάνε στραβά. Και το δεύτερο, όταν κάποιο όπω εσεί κάνει πολύ μεγάλη απαρίθμηση, ε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, ε, να δούμε τι δεν αναφέρατε. Μήπω το είπατε και δεν το κατάλαβα εγώ. Τι θα γίνει, πώ θα θέσουμε τα θεμέλια κατά τη διάρκεια της δική σας προεδρίας ε, να προχωρήσει με τον Καναδά η συμφωνία για την κύρωση. Γιατί πολύ συχνά ολοκληρώνεται ε, μια συμφωνία, υπογράφεται και ε, στη ΣΕΤΑ έχω πολύ μεγάλες ανησυχίες για την καθυστέρηση. Δεύτερο, μιλήσατε για την νομοθεσία και ε, το καθεστώς της Κίνας ε, σε ό,τι αφορά την οικονομία της αγοράς. Κάτι που δεν άκουσα να λέτε ήταν η μεταρρύθμιση του TDI γενικώ. Γιατί το θέμα αυτό με την Κίνα ε, δεν θα λυθεί αν δεν αρθεί η εμπλοκή στο Συμβούλιο για διάφορα μέσα προστασίας του εμπορίου θα σας παρακαλούσα να προσαρμόσετε σχετικά τις προτεραιότητες σας. Τώρα έχουμε τις συμφωνίες ΤΙΣΑ, έτσι που γίνονται διαπραγματεύσεις και στον ΠΟΕ μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι εξελίξεις. Θα μπορούσε να μας υποστηρίξει η Προεδρία να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Επίσης, αναφερθήκατε στη συνεργασία με την Αφρική και σας ευγνωμονώ ιδιαίτερα, γιατί και για μας είναι προτεραιότητα και κέντρο βάρους και θα σας παρακαλούσα πολύ γρήγορα ε, να πιέσουμε για να γίνουν συμφωνίες με τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο και στο Κοινοβούλιο θα προσπαθήσουμε να το πιέσουμε και να το προωθήσουμε αυτό και στο Συμβούλιο παρακαλώ. Θα πρέπει όχι απλώς να συζητάμε την καταπολέμηση των αιτίων της ε, μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και την οικονομική συνεργασία και τι θα κάνουμε το επόμενο εξάμεινο έτσι, σε πρακτικό επίπεδο και αυτό. Και θα σας παρακαλούσα να ξαναδείτε τις προτεραιότητες. Όλες θέλω να τις υποστηρίξω, δεν λέω, αλλά μήπως να τις συμπληρώσουμε κάπως. Ξέρω ότι όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργή να ξημερώσει. Ευχαριστώ. Ο Σχετικά με τι προτεραιότητε, χάρηκα που μιλήσατε για τα ορυκτά. Ξέρω ότι θα πιέσετε όσο μπορείτε κατά τη διάρκεια της προεδρία σα. Χάρηκα επίση που μιλήσατε για την διαφάνεια στο εμπόριο εν γένεια, όπως γνωρίζετε. Από τον Μαυρίκιο πέρασαν πολλά χρόνια για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών προσπαθήσαμε να πιέσουμε για να εγκριθεί η συμφωνία από τα κρατή-μέλη. Είπαμε ότι πέρα από το ότι το θέλουμε, καλό θα ήταν να δώσουμε και το καλό παράδειγμα προς τα έξω. Και επειδή ο Ντανίλ Κασπάρη μίλησε το θέμα. Από το 2001 Ξέρουμε ότι θα τα λέγαμε το 2016, είχαμε ραντεβού αν θέλετε το 2016. Υπήρξε έλλειψη ετοιμότητας από, τα, από τους θεσμούς. Είχατε τόσο χρόνο, πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο ανέτοιμοι πήγαμε στο Ναϊρόμπι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο να μην έχει πάει πρώτα στο Συμβούλιο. Εσείς ως Προεδρία πρέπει να ζητήσετε από την Κομισιόν ε, να έχετε κάτι στα χέρια σας. Πολύ πριν τον Ιούνιο βεβαίως. Αυτό που περιμένουμε και εμείς. Αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο και ο Ντάνιλ έχει δίκιο. Αν ε, θέλουμε να αποφύγουμε την αντιπαράθεση Κοιτάξτε, αν δεν κάνουμε τίποτα ως τον ε, Δεκέμβριο ή δεν κάνουμε την παραχώρηση στην Κίνα θα έχουμε κρίση, θα έχουμε διέξοδο και η λύση θα ήταν να τροποποιήσουμε ενδεχομένω τους αμυντικούς μας μηχανισμούς για να δώσουμε οικονομικό καθεστώς στην ε, Κίνα. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι στο τραπέζι ακόμη λόγω της TDI. Έχουν προχωρήσει τόσες μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν καν είναι αυτό στο τραπέζι του Συμβουλίου. Και ακούμε και νούμερα τα οποία είναι μάλλον ε, υπερβολικά 3,5 εκατομμύρια γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που του οποίους αφορούν τα μέτρα κατά της Κίνας στον τομέα της άμυνας. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι αν δεν αναλάβουμε δράση, επιλούνται πάρα πολλέ θέσει εργασία. Είμαι Μακλάκιν από την ECR. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ για το αισιόδοξο μήνυμα τη Προεδρία. Το θέμα είναι όμω τι τελικώς θα πετύχουμε στο τέλο. Χαίρομαι που θέλετε να προχωρήσετε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, στις Συμφωνίε Εμπορίου. Θέλετε αποτελέσματα και χαίρομαι που ήταν επικοδομητικά ανοιχτή για συνεργασία με το Κοινοβούλιο πάνω στα του εμπορίου. Βεβαίω έχουν ξεκινήσει πολλά πράγματα πριν από εσά. Περιμένω όμω στην ΣΥΤΑ συγκεκριμένα με του Καναδού να σημειωθεί κάποια πρόοδο. Δυστυχώ η Σιγκαπούρη έχει αποκλειστεί κατά τα λοιπά. Ο Καναδά πάντως θα μπορούσε να προχωρήσει αν τηρήσουμε την ατζέντα της άνοιξης. Θα μπορούσαμε ίσως ε, σύντομα να δούμε και την κύρωση. Όσον αφορά τώρα για τα ορυκτά, τα κρίσιμα ορυκτά, ο τριμερής διάλογος ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε του επόμενου 6 μήνε, εκτό αν εσεί πιστεύετε ότι πραγματικά μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η Κομισιόν βλέπω να τροποποιεί τη στάση τη, θα είναι υποχρεωτική, υποχρεωτικό το μέτρο, προαιρετικό. Δεν ξέρω, έχουμε ανάμεικτε εντυπώσει. Πώ θα χειριστείτε το θέμα από εδώ και πέρα του επόμενου 6 μήνε. Και ακόμη και αν αυτό δεν θα κλείσει 6 μήνε, αναφέρατε την Κίνα και την ιδιότητα του κράτους με οικονομία της αγοράς. Πού πήγαινε το Συμβούλιο όσον αφορά αυτό το πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα. Πρέπει σίγουρα πάντως να το συζητήσουμε και κάπου να καταλήξουμε τους επόμενους 6 μήνες. Άλντε. Η κυρία Σχάκα, καλώς την Υπουργέ. Α, θα μιλήσω Ολλανδικά. Ε, που κατα... Ε, αγγλικά που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος και οι Ολλανδοί Υπουργοί. Χαίρομαι για την ευκαιρία που θεωρείτε ότι προσφέρει το εμπόριο για να ενισχυθούν οι κανόνε και το σύστημα. Δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει πάντα ούτε στο Συμβούλιο ούτε στη χώρα μα, παρά τη μακρά ιστορία ανοιχτού εμπορίου που βασίζεται σε αξίε και αρχέ. Και το έχει προωθήσει αυτό το θέμα και η δική μα χώρα. Με περιέργεια περιμένω να ακούσω τι μπορείτε να κάνετε ε, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου για να εξασφαλίσετε ότι όλα τα μέλη του Συμβουλίου θα διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο για να καλυφθεί αυτό το κενό ε, και η απόσταση που μας χωρίζει ε, με τους πολίτες. Το είπατε και εσείς για θέματα εμπορίου, οι πολίτες και όσοι παίρνουν τις αποφάσεις. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά γνωρίζω και από την Κομισιόν, δεν έχουμε συνομιλητή συχνά στο Συμβούλιο για να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα και το χάσμα ε, των λαμβανών της αποφάσεις με τους πολίτες παρόλο που η εντολή ε, έρχεται από τα μέλη του Συμβουλίου. Είπατε ότι ε, θα αντισταθείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα διαφάνειας. Η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, είχε θαυμάσιες πρωτοβουλίες μάλλον η νυν Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξίζει επένου. Γιατί πολύ συχνά ισχύουν στα κράτη-μέλη εθνικοί κανόνε και δυστυχώ στην περίπτωση TTIP δεν είμαστε μόνο εμεί που αποφασίζουμε, υπάρχουν και Αμερικανοί. Τώρα, για ένα άλλο θέμα. Το σύστημα που βασίζεται κανόνες μπορεί να βελτιωθεί με πολλούς τρόπους δεν υπάρχουν μόνο οι διμερείς συμφωνίες αλλά και πολυμερείς διεθνώς. Σήμερα μιλήσαμε για το ε, Ναϊρόμπι αλλά και η συμφωνία για τις ε, υπηρεσίες είναι κάτι που μας απασχολεί και το είπαν οι συνάδελφοι και ε, το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς και η σημασία της Κίνας. Και θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι στην προσέγγισή μας αλλά και νυφάλαιοι με σωστή πληροφόρηση. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εμπόριο εστιάζει στο εμπόριο και τις αξίες. Άρα φαίνεται να παντρεύεται πολύ ωραία με τη δική σας ατζέντα και τις ε, ε, προτάσεις στο Κοινοβούλιο για τα ε, ορυκτά από τις εμπόλεμες περιοχές και τα πασανιστήρια τα είπατε. Θέλω να αναφερθώ λίγο στους στον έλεγχο των εξαγωγών. Εμείς στο Κοινοβούλιο πιέζουμε να έρθουν νέε πρωτοβουλίε. Είναι πάρα πολύ επίγουσα η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμή κάπω αδρανή. Εσεί θα του πιέσετε έτσι ώστε κατά τη διάρκεια τη Ολλανδική Προεδρία να προχωρήσει αυτό το θέμα. Για ένα τελευταίο, ακριβώ όμω επειδή έχει τόσο μεγάλη σημασία για το εμπόριο, συμφωνία σύνδεση με την Ουκρανία. Υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο στα θέματα εμπορίου να ε, παραγωνιστούν ακόμα περισσότερο μετά την πίεση της Ρωσίας. Και κάτι που δεν ενδιαφέρει μόνο τους Ολλανδούς, αλλά πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει δημοψήφισμα στην Ολλανδία κατά πόσο η υπογραφή της κυβέρνησης ε, θα πρέπει να παραμείνει ε, στη Συμφωνία Σύνδεσης με την υποστήριξη της ε, Ολλανδικής Βουλής. Εσείς προβλέπετε ειδικέ πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας ε, για να πείσετε τον κόσμο ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει και να υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ, ο Χέλμουντ Σόλτ. όχι, κυρία Μινουέρ, που είναι και Ολλανδέζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πλόμαν, καλώ ορίσατε. Ε, ήρθατε να μιλήσετε για την Προεδρία σας μαζί μας. Του επόμενου μήνε ξέρουμε ότι είναι οι εξέλιξη στο TTIP, ΣΕΤΑ και ΤΙΣΑ, στις τρεις αυτές συμφωνίες. Να συζητήσουμε λοιπόν τι θα κάνετε με αυτές τις συμφωνίε και ε, τις δεσμεύσεις που αναλάβατε προς το Κοινοβούλιο, ε, που τα κράτη-μέλη ε, υποστήριξαν παρακαλώ ομόφωνα. Τι γίνεται με τα εθνικά κοινοβούλια, προστασία επενδύσεων και δημόσιες υπηρεσίες. Είναι σκληρέ οι διαπραγματεύσει και στη Τίζα και στη ΣΕΤΑ. Την άλλη εβδομάδα στην Τίζα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Ε, η ΣΕΤΑ θα πρέπει να κυρωθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Και στο μεταξύ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έχει και μια απόφαση για το κατά πόσο θα πρέπει το κοινοβούλιο, μάλλον ή, τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις ε, Διαπραγματεύσει για τη Σιγκαπούρη και αυτό θα είναι και προηγούμενο. Μαζί με άλλους 52 βουλευτές έχω υποβάλει μια ερώτηση σχετικά και για το Ολλανδικό Κοινοβούλιο τι θα κάνετε έτσι ώστε να φροντίσετε τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν λόγο για αυτές τις συμφωνίες. Είπατε επίσης ότι θεωρείται απαράδεκτο ότι το ESDS e έχει ε, βγει ε, από το TTIP και όχι από το ΣΕΤΑ, που είναι η επέλυση διαφορών επενδυτή κράτο. Πραγματικά καλά το λέτε, γιατί στο παρασκήνιο γίνονται διάφορες εργασίες και ε, το ξέρουμε ε, και η συμφωνία μιλάει για ένα σύστημα επίλυσης ε, διαφορών σε επενδυτικό δικαστήριο. Ωραίοι εφημισμοί είναι αυτά. Γιατί τα έχετε βάλει στη ε, συμφωνία. Είναι ένα παράλληλο δικαστικό σύστημα πέρα από τη τακτική δικαιοσύνη και τα κανονικά δικαστήρια. Και δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης. Και τους διαιτητές τους πληρώνουμε εμεί. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα και διονύζεται βέβαια κάθε υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρήσουμε ότι το σύστημα ε, δεν γίνεται για να ε, ε, ασκηθεί μια πίεση για να παγώσουν οι ρυθμίσεις. Είναι το λεγόμενο regulatory chill στα αγγλικά. Λοιπόν, παραμένουν να ισχύουν ε, και στο ECS ε, όλες οι ε, διαφωνίες που είχαμε για το ISDS. Η προστασία του επενδυτή δεν θα πρέπει να θίγει ούτε τις προδιαγραφές ούτε τη δημοκρατία μας. Το έχετε διατρανώσει αυτό. τότε γιατί δεν κάνετε κάτι στην κατεύθυνση αυτή και σε δικαστικό επίπεδο εννοώ. Για το TISA αλλά και στο ΣΕΤΑ ισχύει αυτό και στο TTIP, παίζουν σημαντικό ρόλο οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κοινοφελείς και πώς αυτές ορίζονται. Ε, είναι πάρα πολύ σαφής ο ορισμός μιας κοινοφελούς υπηρεσίας. Ε, είναι κάτι, μάλλον όταν κάτι ε, εξ ολοκλήρου χρηματοδοτείται από το κράτος είναι δημόσια υπηρεσία. Στην Ολλανδία αυτό δεν υπάρχει ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε πουθενά και θέλετε να το μεταφέρετε σε 50 χώρες. Ε, ποιες δραστηριότητες εσείς χαρακτηρίζετε δημόσιες υπηρεσίε και κοινοφελή για να μπουν ω εξαίρεση. Στη ε, Ολλανδία αυτό δεν έχει γίνει. Ε, μια τελευταία ερώτηση. Είστε διατεθειμένοι αυτή την στενή ε, έννοια και το στενό ορισμό των δημοσίων υπηρεσιών να το αναθεωρήσετε. Να ορίζουν δηλαδή οι κρατικές αρχές και τοπική αυτοδιοίκηση τι εστί δημόσια και κοινοφιλής υπηρεσία και να κανονίζουν την πορεία σας. Ο Γιάννη Ζαντό από τους Πρασίνους. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που ήρθατε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ορυκτών από εμπόλεμες περιοχές, συγκρούσεων, τα αιματοβαμμένα ορυκτά. Είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο. Αναφέρατε κι εσείς τους πληθυσμούς που είναι θύματα εκμετάλλευσης, ε, μορφών βίας και ένα σωρό άλλων αφρικαλαιοτήτων εξαιτία των ορυκτών αυτών. Ε, δεν θα συζητήσω την καλή πίστη και την καλή βούληση των όσων παρευρέθηκαν στον Ταβός, αλλά το θέμα που βρίσκεται επιτάπητος είναι λίγο πιο πιεστικό. Μέσα στα πλαίσια της due diligence, όπως λέμε, πρέπει να ε, εξεταστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, τη δέουσα επιμέλεια. Ε, θα πρέπει λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί εδώ μια αξιόπιστη λύση σε επίπεδο Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου δεν σας διαφεύγει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν, αποφάσισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία με το Μαρόκο, συμπεριλαμβάνοντας το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Είναι θέμα διεθνών συνθήκων. Και το Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα, θα προσβάλλει την απόφαση αυτή, που για άλλη μια φορά θα μας φέρει σε παράβαση και σε παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Βάσει ποιων αρχών τα μαροκινά προϊόντα φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ως προς τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Το ίδιο και πάλι. Εφόσον δεν έχουμε ακόμη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου για το καθεστώς της Συμφωνίας με τη Σιγκαπούρη, εάν θέλετε σκέφτεστε να υπογράψετε τη συμφωνία με τον Καναδά, βάσει ποια νομικ... με ποια νομική βάση θα το κάνετε. Και σε ό,τι αφορά τι διατλαντικέ διαπραγματεύσει, το TTIP και όλα τα σχετικά. Μιλήσατε για διαφάνεια. Πολύ ωραία. Αν ακούσω όμω τα όσα είπατε για τη διαφάνεια, θα θεωρήσω ότι περισσότερο ε, έχουμε μια περίπτωση επικοινωνιακή πολιτική μεταξύ θεσμικών οργάνων. Είναι λίγο προπαγανδιστικά όσο μα λέτε. Δηλαδή, θέλετε ε, μια γλώσσα εύληπτη για όλου του Ευρωπαίου για να καταλάβουν όλα τα ωφέλη αυτών των συμφωνίων συμφωνιών. Δηλαδή, εάν ευθύ εξ αρχή λέτε ότι μόνο ωφέλη έχουμε να αποκομίσουμε από μια τέτοια συμφωνία, δεν λέγεται αυτό διαφάνεια, προπαγάνδα λέγεται. Για μένα, διαφάνεια στι διαπραγματεύσει αυτέ θα ήταν λόγου χάρη όταν βρίσκεστε στη Χάκη να μπορείτε να δείτε το διαπραγματευτικό έγγραφο μπροστά σα, στο γραφείο σα και όχι ε, μόνο όταν έχετε τον πρέσβη των ΗΠΑ. Οι συνδικαλιστικέ οργανώσει, οι πολίτε, οι ενώσει καταναλωτών εκεί θέλουν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων. Όχι μόνο οι βουλευτέ που μπορεί να έχουν στίβε εκατοντάδων σελίδων, χωρί να έχουν μια ομάδα συνεργατών για να μπορέσουν να πείσουν νομικώ τι σημαίνουν όλα αυτά. Ε, επί τη ουσία λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τη διαφάνειά σα νομίζω και ο τρόπο που προσεγγίζεται το όλο θέμα ενώπιον τη κοινή γνώμη, τι εμπορικέ διαπραγματεύσει, δημιουργεί περισσότερη καχυποψία παρά επιλύει προβλήματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν μελέτε που λένε ότι η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση και, άλλοι που άλλε που λένε ότι θα τι καταστρέψει. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αποσχολεί του Ευρωπαίου πολίτε και δεν είναι απλώ επικοινωνία τέχνασμα να προσπαθήσουμε να του πείσουμε ότι η συμφωνία αυτή θα έχει ωφέλη. Ευχαριστώ από την EFTT. Η κυρία Πεκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ενώσω τη φωνή μου στα καλωσορίσματα των συναδέλφων προς την Επίτροπο μάλλον συγγνώμη την Υπουργό, την ευχαριστώ που μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας. Άκουσα την παρουσίασή σας μεγάλη προσοχή και διάβασα και το έγγραφο με το πρόγραμμά σας. Τώρα, για το καυτό ζήτημα που έθιξε και ο τελευταίος ομιλητής, ο κ. Ζαντό, να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μου ως προς τις διαπραγματεύσεις ε, της συμφωνίας TTIP και κάποιες δηλώσεις σας που δείχνουν ε, την διάθεση να υπάρξει επιτάχυνση για να μην πω και ολοκλήρωση των ε, διαπραγματεύσεων αυτών επί της θητείας του κ. Ομπάμα. Επ' αυτού να σας κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για λίγο, γιατί θα θέλαμε αυτή η βιασύνη να μην προκαλέσει και παράδεκτους συμβιβασμού. Ακόμη απέχουμε πολύ από μια τελική συμφωνία σε θέσεις για τα επιμέρους κεφάλαια, όπως για τις γεωγραφικές ενδείξεις ή τις δημόσιες προμήθειες, που δεν φαίνεται να οδηγούν σε κάποια λύση. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα TTIP ε, μεσοβέζικο, ε, ούτε να δοθεί μία ε, πλήρης εκχώρηση αρμοδοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Κοινοβούλιο. Θα σας παρότρινα λοιπόν να αντιταχθείτε σε κάθε τέτοιου είδους λύσεις. Ένα άλλο επιχείρημα που επίσης πολλοί έθιξαν είναι η αναγνώριση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς για την Κίνα. Και σε αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνω ότι για μας είναι σημαντικό και σοβαρό να συζητηθεί το θέμα και στο επίπεδο του Συμβουλίου ακόμη. Να μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με την εξισορρόπηση διαφορετικών συμφερόντων. Σκεφτείτε λοιπόν τις συνέπειες ή ασδήποτε αποφασή σας για όλον μας τον εμπορικό κλάδο και τις βιομηχανίες μας. Και τέλος, ένα άλλο θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλές, δηλαδή τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, τα ορυκτά των συγκρούσεων, ένα θέμα που λέτε ότι θα εξετάσετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη το εξή. Είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ακόμη και αν υπάρχουν πολλές μεταβολές, πιστεύω ότι όσο έχουμε αυτή την αγορά στα χέρια μας, μην χάσουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Αναθέτω λοιπόν τις ελπίδες μου στην, ε, στον κοινό νου και τη λογική όλων. Κύριε Αλεπένα Λεπέν από την ομάδα της. Ναι. Κύριε Υπουργέ. Έχασα την αρχή της ε, μιλής σας. το κύριο πρόβλημα, πρόβλημά μας είναι η σταθερότητα, η, η αστάθεια μάλλον που προκαλούν οι εξτρεμισμοί και ξαφνικά νομίζω ότι μιλάγατε για τον ΤΑΕΣ, για τους τρομοκράτες, τους τζιγαντιστές και μετά μιλούσατε για πολιτικές δυνάμεις που απλώ διαφωνούν με τις πολιτικές σας προτιμήσεις. Υπάρχει πρόβλημα με τη διαφάνεια που επικαλείστε και την έκθεση για τη δημοκρατία και τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών. Και καταλήγω ότι μέσω ημών, με η Προεδρία θεωρεί ότι πρέπει οι άλλοι να καταδικαστούν στο του εξωτερών ως εξτρεμιστές. Δεν υπήρχε το πρόκειται. Ε, μα κοιτάξτε, προφανώς κάποιοι θα διαφωνήσουν. Έχετε πολύ σημαντικά θέματα μπροστά σας. Κάποιοι θα διαφωνήσουν, εννοείται. Την τεράστια κρίση των μεταναστών, την τρομοκρατία, την καταργήση του Σέγγεν, την ε, των Άγγλων που θέλουν να βγουν από την Ένωση. Αυτά βεβαίως είναι τεράστια προβλήματα, είναι εν πάση περιπτώσει θέματα τα οποία η Ολλανδική Προεδρία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Δεν έχω καμία αμβολία, θα κάνετε βέβαια τα ίδια με τους προηγουμένους. Εν πάση περιπτώσει να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν θίξατε, που είναι η κατάσταση στη Γεωργία. Και δει, στη Γεωργία, στη χώρα μου, η Ευρωπαϊκή Αγροτική Αγορά, χάρη στην Κομισιόν, τη καλέ τη υπηρεσίε, έγινε υπερανταγωνιστική. Σε εμά κάθε δύο μέρες ένας αγρότης αυτοκτονεί προσπαθώντας να κάνουν τα αγροκτήματά τους ε, πιο ανταγωνιστικά. Και όμως απελπίζονται γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Κλείνουν επιχειρήσει μία με την άλλη. Και το λέω αυτό στην την προσοχή των Γάλλων και των άλλων Ευρωπαίων. Το Κοινοβουλίο, η Κομισιόν είναι συνυπεύθυνοι γιατί τροποποίησαν θεμελιωδώς την φιλοσοφία τη γεωργίας και την έκαναν μια αγορά σαν όλε τι άλλε. Οπότε το ερώτημα το οποίο θέλω να σα θέσω είναι θα ασχοληθεί καθόλου με το πρόβλημα ή θα κάνετε τα ίδια με του προηγούμενου. Θα υπογράψετε με την Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, με μεγάλου παραγωγού συμφωνίε την στιγμή που αυτοί παράγουν κρέας πολύ φθηνότερο από το δικό μας για να μην μείνει τίποτα από την γαλλική κτηνοτροφία. Ένα θεμελιώδες ερώτημα λοιπόν. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα πραγματικά μελήματα των λαών της Ευρώπης, των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ περισσότερο από την πολιτική επιχειρηματολογία που προσπαθήσατε να αναπτύξετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, συνάδελφοι, έχουμε τώρα το εξής πρόβλημα. Κάθε πολιτική ομάδα ζήτησε ε, μάλλον έκανε τουλάχιστον τρεις ερωτήσεις και ο χρόνος μας τελείωσε, άρα δεν μπορούν να μιλήσουν άλλοι συνάδελφοι. Κατάλαβατε τι έγινε τώρα. Ίσως οι πολιτικές ομάδες να το συζητήσουν αυτό στο ιστορικό τους το πρόβλημα για να βρουν και άλλες λύσεις. Για να μπορούν να μιλούν και άλλοι βουλευτές και να κάνουν ερωτήσεις τέτοιες. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει. Δέκα λεπτά να απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις που κάνατε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα σχόλιά σας σε τρεις γύρους. Τον αφορά τα, τον πολυμερή χαρακτήρα, θα είμαι σύντομη ως προς αυτό. Τα, έχετε, τα με την Επίτροπο για την ΣΥΤΑ, την TTIP, αλλά και την Γεωργία και το θέμα το νομοθετικό. Ακούγοντας τα σχόλιά σας, Πιστεύω ότι πρέπει να πω ότι βεβαίω είναι η πρώτη φορά που συναντώμεθα και είναι φυσικό να υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις διάφορες προτεραιότητες. Αν ξέρετε πάντως πόσο ελεύθερη, πόσο ανοιχτή είναι η Ολλανδία όσον αφορά τις ε, ελεύθερες συναλλαγές και πώς Βεβαίω στηρίζουμε και τα θέματα βοήθεια και πώ προσπαθούμε να τα συγκεράσουμε σε όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε, δεν υπήρχε τελικά άλλη επιλογή. Με αυτά τα θέματα πρέπει να ασχοληθούμε. Αυτά είναι τα θέματα, αν και κάποιοι κατέθεσαν και άλλα θέματα στο τραπέζι, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Γι' αυτό είπα, θα είμαστε εδώ και θα δουλεύουμε νυχθημερών. Πώ προσεγγίζουμε όμω το εμπόριο και είμαστε πραγματικά ανοιχτοί. Πιστεύω ότι, όπω προείπα, δεν είμαστε δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά, γι' αυτό να πω δύο λόγια. Όταν μιλάμε για το εμπόριο και τις εμπορικές συμφωνίες, να μην έχουμε μόνο τη μία πλευρά, τη μία ομάδα, τη μία φωνή, να αφουγκραστούμε όλες τις πλευρές. Εγώ μίλησα με οικονομολόγους όπως Στίγλιτς, ο Καπάλτο και την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, τον Γκάσφαν Χάρτεν και μιλήσαμε για το πώς βλέπει το διεθνές σύστημα δικαστηρίων, το σύστημα των διεθνών δικαστηρίων. Μίλησα όμω και με ΜΚΟ και με επιχειρήσει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι η πραγματική διαφάνεια. Όχι να συνεχίζει κανείς να κάνει αυτό το οποίο νομίζει ότι είναι το σωστό, αλλά να ακούει τους πάντες και να προσπαθεί να ενσωματώσει τις διστάμενες απόψει και να καταλήγει σε μία πρόταση. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας έτσι θα προχωρήσουμε. Καταρχήν για την ΤΙΣΑ τη συμφωνία τη συναλλαγή των τομέα υπηρεσιών, την οποία ανέφεραν πολλοί από εσά. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εισηγήτρια, την κυρία Vivian Ρέντινγκ, διότι η ίδια και εσεί επιτελέσατε πολύ σημαντικό έργο στην επίτευξη συμβαστικών τροπολογιών που συγκεράζουν τι απόψει του πολιτικού φάσματος εν το συνόλο του. Ευχαριστώ πολύ για το έργο σας λοιπόν. Τώρα για τις κοινοφελείς υπηρεσίε. Φυσικά θα τύχουν προστασίες. Η ΤΙΣΑ δεν θα ζητά από τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιήσουν οποιαδήποτε υπηρεσία κοινή ωφέλεια, ούτε θα αποτρέπει, ούτε θα απαγορεύει στις κυβερνήσεις να επεκτείνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κατάλογος. Ο οποιοδήποτε κατάλογος ήταν περιοριστικός στο πλαίσιο της ΤΙΣΑ δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις κυβερνήσεις. Θέλουμε οι κυβερνήσεις να ορίζουν τι είναι κοινή ωφέλεια και να μπορούν να τροποποιούν τη στάση τους από καιρούς καιρών. Δεν θέλουμε λοιπόν κατάλογο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ανησυχείτε. Φυσικά είναι θεμητό να ανησυχεί κανείς, όμως ε, πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο προχωράει η συμφωνία πρέπει να είναι καθυσιαστικό για του περισσότερου. Συμφωνούμε λοιπόν επ' αυτού. Για την TTIP τώρα, την Διατλαντική Συμφωνία, κατανοώ ότι και συμφωνώ με αυτού που είπαν ότι μια καλή συμφωνία είναι πολύ πιο σημαντική από το να πετύχουμε μια οποιαδήποτε συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν, βιαστικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ όμω, για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, να το κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Φυσικά υπάρχουν πολλά ζητήματα που εκκρεμούν. Γνωρίζετε ότι έχουμε μπροστά μας διαφορούς γύρους διαπραγματεύσεων. Κάποιοι από αυτούς θα γίνουν τους επόμενους έξι μήνες. Συμφωνώ όμως ότι μια κακή συμφωνία δεν είναι συμφωνία για μας. Μίλησα για την ενημέρωση του κοινού προηγουμένως και είπα ότι είναι σημαντικό να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θα είμαστε επιθετικοί στην ενημέρωση του κοινού, συμφωνώ με την πρακτική αυτή και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και την Επίτροπο που υποστηρίζει αυτήν την κατεύθυνση. Όσον αφορά την ΣΥΤΑ, τη συμφωνία με τον Καναδά, την ανέφερα εν συντομία, ευχαριστώ που την αναφέρετε. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τους νομικούς, είναι πάντως μια πολύ σημαντική συμφωνία, εννοείται, και θα θέλαμε να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν. Αναγνωρίζουμε ότι στην ΣΥΤΑ οι διατάξει για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση των διαφορών τροποποιήθηκαν, εξυγχρονίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τώρα οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες στην ΣΥΤΑ για να ευθυγραμμιστούν με τις τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα όπως αυτές που έχουν προτείνει και στο πλαίσιο της TTIP. Έχουμε διαπραγματεύσεις που τρέχουν με την νέα Καναδική κυβέρνηση και γι' αυτόν τον λόγο ίσως χρειαστεί λίγος περισσότερος χρόνος για να καταλήξουμε. Διότι είχαμε εκλογέ. Στον Καναδά άλλαξε η κυβέρνηση και άλλαξε και λίγο η στάση του Καναδά. Και φυσικά χρειάζεται και η νέα καναδική κυβέρνηση λίγο χρόνο για να εξετάσει το θέμα. Οι συνομιλίες λοιπόν συνεχίζονται και νομίζω ότι είμαστε κοντά στην επιτευξή συμφωνίας. Επίσης, όσον αφορά την Ιαπωνία, η πρόοδος εκεί ήταν απογοητευτικά αργή. Το είπατε μερικοί από εσά. Και εδώ, ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει ότι θα θυσιάσουμε το περιεχόμενο. Και εδώ πιστεύω θα καταλήξουμε σε κάποια καλή συμφωνία, φιλόδοξη συμφωνία σε όλους τους τομείς. Να είμαστε όμως ρεαλιστές. Γιατί έχουμε και την TPP, Συμφωνία είπα Καναδά Ασίας, κάποιες έννοιες, κάποιες διατάξεις της TPP εμπνέονται από διατάξεις της TTIP κάτι το οποίο δεν κάνει ευκολότερες τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία και την Mercosur. Ξέρω ότι τα ανακατεύσα λίγο με τις προτεραιότητες αλλά αυτό είναι και στην ατζέντα της δικής σας επιτροπής. Λοιπόν, οι σχέσεις μας με την Λατινική Αμερική είναι πολύ σημαντικές και στην περιοχή αυτή συνέβησαν αλλαγές, έχουμε νέες κυβερνήσεις, ε, δύο χώρες. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι υπέρ των συνομιλιών. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τις επόμενες, τους να σημειωθεί πρόοδος αφού γραζόμενοι βεβαίως όλες τις ανησυχίες στο Συμβούλιο και αλλού. Θα είμαστε και εκεί όμως αμυντικοί αλλά και επιθετικοί αν θέλετε όπου χρειάζεται όσον αφορά τις EPA. Όπως είπα, υποστηρίζουμε αυτές τις συμφωνίες στην Δυτική Αφρική έχουμε μια ευκαιρία να τους βοηθήσουμε να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονώντας τις επενδύσεις, τονώντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας τις παραγωγικές τους δυνατότητες. Θα προωθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεχιστούν επικοδομητικά συνομιλίες με τις χώρες αυτές της Δυτικής Αφρικής ε, είμαστε θεωρώ ένας έντιμος διαμεσολαβητής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των χωρών της Δυτικής Αφρικής. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό οικονομία της αγοράς, πολλοί από εσάς συμφωνούν ότι πρόκειται για προτεραιότητα. Είναι μια σημαντική προτεραιότητα Πρόκειται και για ένα ζήτημα το οποίο θα επηρεάσει πολλούς από εμάς. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι θα επηρεαστούν άνθρωποι ή θέσει εργασία ιδιαίτερα στο υψηλότερο επίπεδο, στις υψηλότερες αμοιβέ, αλλά μια θέση εργασία είναι μια θέση εργασία. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το θέμα. Έχει σχέση με την αμυντική μας στάση στον τομέα του εμπορίου. Θα γίνει ένας ποτός γύρω συζητήσεων για, την, τον χαρακτηρισμό οικονομίας της αγοράς κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας και θα πιέσουμε την Κομισιόν. Συμφωνώ με πολλούς από εσάς που είπαν ότι έχει λιμνάσει το θέμα για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε λοιπόν συζητήσεις στο Συμβούλιο. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να βασίζονται, να περιστρέφονται γύρω από μια πρόταση της Κομισιόν. Θα εξετάσουμε την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο, την πρόταση της Κομισιόν εννοώ, με επικοδομητικό πνεύμα και με στόχο βεβαίω το να καταλήξουμε σε κοινή θέση το συντομότερο δυνατόν. Και εδώ θα ενθαρρύνουμε την Κομισιόν, να το πω διπλωματικά για να μην πω θα την πιέσουμε, να υποβάλει πρόταση, να καταθέσει πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Όσον αφορά τη σύμβαση και τη διαφάνεια, την αναφέρατε κι εσείς. ότι μετά από τον μπλοκάρισμα των Ευρύτου του 2014 ε, γνώμε, δίστανται μεταξύ των κρατών μελών επί της ουσίας της πρότασης της Κομισιόν. Εμείς ως Προεδρία δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ότι η το στο Συμβούλιο δεν αφήνει περιθώριο εξέβρεσης κοινή λύση λόγω δύο δισταμένων προτάσεων. Η Κομισιόν όμω επέστρεψε να θεώρησε, επανεξέτασε την πρότασή της για τους μηχανισμούς κρατικών προμηθειών και υποσχέθηκε να υποβάλει νέα πρόταση, γνωρίζοντα βεβαίω την θέση του Συμβουλίου. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη στο Συμβούλιο, αλλά είναι μάλλον υπερβολικά νωρί να πούμε οτιδήποτε σχετικά με το αποτέλεσμα. Για την σύμβαση λοιπόν για την διαφάνεια εξετάζουμε δίμερος το θέμα και εδώ έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να δούμε λοιπόν που θα μπορούσαν να εξελιχθούν κάποιες ε, διαφωνίες. Θεωρούμε πάντως ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο για την υπογραφή συμφωνίας. Ακόμη τουλάχιστον. Να ξέρετε όμως ότι εμείς ως Προεδρία και το λέω προς τους εξαριστερών μου θα συνεχίσει να εργάζεται και θα δει το θέμα διμερός ώστε ενδεχομένως η επόμενη Προεδρία να μπορέσει να καταλήξει συμφωνία. Για τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες εξετάζουμε το θέμα από το φως των τροπολογιών που έχετε καταθέσει από 20 Μαΐου. Στις 18 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο έρθει στην Προεδρία να διαχειριστεί τις διαπραγματεύσεις όπως είπα και στην εισήγησή μου στην εισαγωγή μου. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια πρόταση για, τον, την εθελοντική προσέγγιση και υπάρχει πρόταση για ένα υποχρεωτικό σύστημα. Εδώ, ξέρετε, θα σας καλούσα όλους να μην δείτε αυτές τις δύο λύσεις ως ε, αμοιβαίως αποκλειόμενες. Μπορούν να συγκεραστούν. Στην Ολλανδία ξέρετε ότι είχαμε ανέκαθεν συμμαχικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις συνασπισμού. Αυτό ισχύει και σήμερα. Και μέσα σε ένα συνασπισμό καταφέρουμε ακριβώς αυτό, να συγκεράζουμε διστάμενες απόψεις. Αυτό μπορεί να γίνει. Όχι μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι πολλοί συμμερίζονται αυτήν την θέση την αξία της εργασίας δηλαδή και είμαι βέβαιος, βέβαια, ότι θα μπορέσουμε να συγκεράσουμε τις δύο προτάσεις. Εγώ προσωπικώς θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, στη συμφωνία. Όχι μόνο γιατί είναι σημαντικό για εμάς, αλλά διότι είναι ένα σημαντικό θέμα για εκείνους, για τους ανθρώπους που παράγουν τμήματα των κινητών τηλεφώνων, των iPhones που όλοι χρησιμοποιούμε. Τώρα για τον κανονισμό κρατών βασανιστήριων. Να προσθέσω σε αυτά τα οποία ήδη είπα ότι γνωρίζουμε τις ελλείψεις που έχουν όλες οι προτάσεις στο τραπέζι, όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε τις ελλείψεις μέσω του διαλόγου. Εννοείται ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας για να καταλήξουμε και εδώ σε αποτέλεσμα. Κάθε φορά που συζητούμε διμερός με τους ε, διάφορους εμπλεκόμενους, τους βασικούς εμπλεκόμενους. Όσον αφορά την Ουκρανία και τη σχετική συζήτηση και την ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία, Μία διάσκεψη που έχουμε ήδη σχεδιάσει, προγραμματίσει, είναι στα μέσα Μαρτίου. Εγώ θα πάω στην Ουκρανία υπό την ιδιότητά μου της Ολλανδής Υπουργού μαζί με Ολλανδική Αντιπροσωπεία, Εμπορική Αντιπροσωπεία στην Ουκρανία και θα μιλήσουμε κυρίως για γεωργία, για, για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και θα μιλήσουμε εκεί με επιχειρηματίες καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. Η συμφωνία αυτή είναι κατεξοχήν ευκαιρία για την Ουκρανία να εξυγχρονίσει την οικονομία της, να αναπτύξει την δημοκρατία της. Και η δημοκρατία σημαίνει να ακούγονται όλες οι φωνές. Σημαίνει κράτος δικαίου. Πράγματα τα οποία βεβαίω υποστηρίζουμε μέσω της συμφωνίας. Διότι υποστηρίζουμε κάθε ευκαιρία που έχουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Μετανάστευση. Βεβαίως είναι βασική μας προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για διάφορα συμβουλία, για διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου. Η Επιτροπή σας, αλλά και η Επιτροπή Ανάπτυξης, με την οποία μιλάω αναγνωρίζει την σημασία κάποιου ολοκληρωμένου πακέτου δέσμης μέτρων για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν την κρίση των μεταναστών και των προσφύγων. Λίβανος και η Ορδανία προκειμένου. Ο Λίβανος πέρα από το πακέτο πρέπει να υποφεληθεί και των εμπορικών μέτρων. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τι χώρε αυτέ λοιπόν με τέτοιου είδου προτάσει, στον τομέα του εμπορίου. Έτσι επενδύουμε σε, με τρόπο δομικό στην οικονομική ανάπτυξη. Ενισχύουμε δηλαδή τι χώρε και το ρόλο του στην περιοχή. Χώρε που κάνουν παραπάνω από όσο αναλογεί στην υποδοχή προσφύγων. Καθώς ενώ λοιπόν περιμένουμε και λύση στο συριακό πρόβλημα. Εν κατακλείδη, τέσσερα θέματα, πολύ σύντομα όμως. Θα σας αποκαλώ σέρα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εξονισμός TDI. Και ο Κασπάρη είπε κάτι. Η πρόταση έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, για να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε ενδεχομένω νέα πρόταση από την Κομισιόν. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, θα το δούμε. Πάντω, μόλι την έχουμε, θα κοιτάξουμε να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αν και αυτό μπορεί να σχετιστεί με την Κίνα και τον χαρακτηρισμό τη οικονομία τη αγορά, Γιατί και εκεί περιμένουμε πρόταση τη Κομισιόν, όπω γνωρίζετε. Κυρία Σχάκε, είπατε για τον έλεγχο των εξαγών. Καταλαβαίνω πόσο πιεστικό είναι το ζήτημα. Και εδώ πιέζουμε να προχωρήσει ο φάκελο με το που θα καταθέσει φυσικά η Κομισιόν τη σχετική πρόταση. Σύντομα ελπίζω. Κύριε εδώ για τη συμφωνία με το Μαρόκο. Η απόφαση του δικαστήριου είναι πολύ πρόσφατη, όπως γνωρίζετε. Πρέπει να τη μελετήσουμε πολύ προσεκτικά πριν κάνουμε τα επόμενα βήματα. Τώρα, η γεωργία είναι προφανώς πολύ μεγάλη σημασία στο μέσο, όχι μόνο για την Γαλλία ή τα κρατημέλη εν γέννη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Το 2050 θα πρέπει να ταΐζουμε 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους και πρέπει να διασφαλίσουμε τότε ότι η γεωργία δεν ενδιαφέρει μόνο τις μεγάλες πολυεθνικές, αλλά και τους μικρού, μικρούς γεωργούς. Αυτά τα συμφέροντα πρέπει να συγκεράσουμε. Πάντως το ελεύθερο εμπόριο είναι μια τέλεια ευκαιρία για την γεωργία. Το έχουμε αποδείξει εμείς. Έχουμε, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγής γεωργικών προϊόντων στον κόσμο. Θαυμάσια! Υπέροχα, σας ευχαριστώ πολύ Υπουργέ και σας ευχαριστώ και πάλι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και εδώ στην Επιτροπή μας. Δεν είναι η τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο καλό να πάτε. Okay, dear colleagues. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Dann kommen wir zu Ερχόμαστε. Punkt 6 der ersten Abstimmung. Σημείο 6 είναι η πρώτη ψηφοφορία. Um sicherzugehen, dass alles seinen richtigen Weg geht. Λοιπόν, για να γίνουν όλα σωστά, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε όλοι μαζί σας ε, τις κάρτες για να αρχίσει η ψηφοφορία. Und die Πέρας ψηφοφορίας. 37 anwesend. 37 παρόντες, 34 ε, ψήφισαν. Ωραία, πάμε στο σημείο 6 λοιπόν να ψηφίσουμε. Ε, είναι αναδιατύπωση ε, των ρυθμίσεων για τα προϊόντα προέλευσης ορισμένων χωρών ΑΚΕ. Έχουμε πρώτα μια ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο της έκθεσης ψηφιπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και το νομοθετικό ψήφισμα ηλεκτρονικά θα το ψηφίσουμε αυτό παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία 34 υπέρ εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Στον κύριο Βαλέσα, τον εισηγητή. Πάμε στο σημείο 7 τώρα. Η θέσπιση εκτάκτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη δημοκρατία της Τινησίας. 52 είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και μία είναι η συμβιβαστική Δεν θέλω να επηρεάσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, να σας πω ότι η συμβαστική τροπολογία υποστηρίζεται και εγκρίνεται και από τα άλλα θεσμικά όργανα. Αν περάσει μόνο αυτή η συμβαστική τροπολογία, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τριμερείς διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο και θα περάσει ως έχει η απόφαση γιατί την εγκρίνουν και τα άλλα θεσμικά όργανα, χωρίς να θέλω να σας επηρεάσω. Παρ' όλα αυτά, φυσικά θα ψηφίσουμε με τη σειρά άλλες τροπολογίες και πάμε. Η τροπολογία τώρα υπαριθμών 1 και δύο είναι για απόρριψη, ψήφι Είναι δύο τροπολογίες για απόρριψη. Κατά αποχές απορρίπτονται οι τροπολογίες που ζητούν απόρριψη. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 6. ψηφιπέ, Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε. Η τροπολογία υπαριθμών 7. ψηφιπέ, Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός. Στην 7 τροπολογία αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Την τροπολογία παρθμών 9. Ναι. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 11 υπέρ. Κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 11 παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 12 και 13 μαζί είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία άκρη 3 υπέρ. Σε επί είναι κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την τρία της άγκρη αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παρελθόν 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παρελθόν 16 υπέρ κατά άποχες. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά χρειάζεται έλεγχο αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Έχει απορριφθεί όντω. Τροπολογία παρελθόν 17 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 19 είπε Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά χρειάζεται έλεγχο και πάλι. Για την 19 κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η άγκρη 6 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 ψήφι υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 20 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 22 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία παριθμό 23 ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται 24 και 25 μαζί Ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 26 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία περιθμών 28 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία περιθμών 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία περιθμών 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία περιθμών 33 υπέρ Τσεκ. Α, για την 31. καλώ. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τροπολογία 31. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 33. Ψήφι φυπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 29 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 35 τσεκ θέλετε ας την ελέγξουμε 29 λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα πέρας Απορρίψετε. Η τροπολογία υπαριθμών 35. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 36. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 37. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ή 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία παριθμών 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία παριθμών 41 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 41 αρχίζει τώρα Πέρας. Απορρίπτεται. 40 ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 50 έχει αποσυρθεί. Και πάμε στην τροπολογία 42 ψηφιπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 43 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, αρχής ψηφοφορία τώρα. Πέρας. Να απορρίπτεται. Η 47 ψήφι υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται η 44 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται η τροπολογία 45 ψηφιπέ κατά άποχες απορρίπτεται η τροπολογία 46 έλεγχο θέλετε για τη 45 ελέγχουμε λοιπόν τη 45 ηλεκτρονικά αρχίζει η Πέρας. Η τροπολογία 46. Υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 48 Υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 49 ψήφι Κατά. Έλεγχος. Για τη 49. Λοιπόν, την επαληθεύουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ισοψηφία απορρίπτεται. Η τροπολογία 52. Ψήφι κατά άποχες και αυτό θέλει έλεγχο λοιπόν 52 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται η τροπολογία παριθμό 51 ψήφι κατά άποχες απορρίπτεται και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί, αλλά α το ελέγξουμε ξανά. Ε, το κείμενο της Κομισιόν όπω τροποποιήθηκε αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, κοιτάξτε, οι πράσινοι είστε υπεράριθμοι. Ε, πέρας. Μάλλον όχι, ψηφίσαν περισσότεροι υπέρ από όσους είχα δει προηγουμένως. Λοιπόν και το νομοθετικό ψήφισμα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ντεσσαρνέ. Yeah, Η κυρία Δεσσαρνές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν ε, μικρή η διαφορά, ε, περίπλοκο το αποτέλεσμα και το να βρούμε ισορροπία, αλλά ελπίζω να επιβεβαιωθεί και στην Ολομέλεια και να ευχαριστήσω τον καθέναν και την καθεμιά από τους συναδέλφους, διότι είναι για αυτούς ευαίσθητο θέμα στην κάθε χώρα. Ακριβώς το θέμα του ελαιόλαδου η συμφωνία προβλέπει ότι αν εντό ενό έτου διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ε, προβλέψει μέτρα για να διορθώσει την έλλειψη ισορροπία εφόσον υπάρχει. Να προσθέσω κάτι. Τη στιγμή που την Ισία αντιμετωπίζει φοβερότατε δυσκολίε, σοβαρότατε ε, δυσκολίε. η Επιτροπή μα επιτέλου αποστέλει ένα θετικό μήνυμα το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό τη Τινησίας στο πλευρό των Τινήσεων και προτείνουμε να εκφράσουμε την ελληνική μας χειροπιαστά, ρεαλιστικά ε, και στην ε, πράξη με, σε συνεργασία με τις θυνησιακές αρχές. Σας ευχαριστώ λοιπόν, λοιπόν πολύ για αυτήν την στάση που είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή και για την νησία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δησανές. Λοιπόν, και ακολουθεί το επόμενο σημείο παριθμών 9 στην ημέρη σε διάταξη που είναι το ψήφισμα για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία μαζί και έχουμε τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 πρώτη. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 του κυρίου Γιάννικ Ζαντό. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται η συμβαστική 3 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική παριθμόν 4 ψήφι υπέρ κατά Enthaltungen. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Dann kommen wir... Και στη συνέχεια έχουμε την τροπολογία υπάρχουν 39 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία τσεκ αλλά ας ελέγξουμε τι 39, αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 42 λοιπόν ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 43. 43 ψήφι Ταγκή. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 6 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 46 ψηφιπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 48 όχι καταπίπτει. Συμβαστική 7 ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 53 ψήφι υπέρ, κατά, άποχες, έλεγχος χρειάζεται εδώ για την 53, αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Η συμβαστική παριθμών 8 Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμό 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συγχαρητήρια για Νίκ. Η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Το δεύτερο τμήμα αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε η συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές έλεγχο θέλει εδώ αρχίζει ψηφοφορία πέρας απερίφθη με μία ψήφο διαφορά και 20 αποχές παρακαλώ η 12 συμβαστική υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 12 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολόγια παρελθόν 2 ψηφιπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε την ούτως τροποποιηθή σε πρόταση ψηφίσματος αρχίζει ψηφοφορία τώρα και λίγοι μέσους 32 υπέρ εγκρίνεται. Πρόεδρε, συγγνώμη, κυρία Σχάκε, ένα διαδικαστικό. Κάνει 3.000 βαθμούς εδώ πέρα, δεν αντέχω, θα σκάσω από τη ζέστη και φαντάζομαι δεν είμαι η μόνη. Τουλάχιστον αφήσουμε την, πρώτα, την πόρτα ανοιχτή και να δούμε τι τρέχει. Γιατί πραγματικά δεν αισθάνομαι καλά και θέλω να ψηφίσω, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει τρομερή ζέστη μέσα στην αίθουσα. Ναι, κατανοώ πολύ τους Μαρίτσι αυτό που λες. Θα ζητήσαμε να αλλάξουμε αίθουσα, ε, να αλλάξουμε και θερμοκρασία εδώ. Ας αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 10 τώρα. Πάει η ψηφοφορία, τελείωσε. Όχι, έχουμε να ψηφίσουμε το θέμα της οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Δυτική Αφρική, εξέταση ερώτησης. Μία ε, μοναδική ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. Με 35 ψήφους εγκρίθηκε και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα τελειώνουν οι ψηφοφορίες σε αυτό ακριβώς το σημείο και πάμε στο 11. Στο 11 η κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος θέλει να φύγει τώρα παρακαλώ ε, σιωπηρός. Έχουμε αυτόν τον καιρό δύο τριμερείς διαλόγους εν εξελίξη. Το πρώτο έχει να κάνει με τα βασανιστήρια και την αντίστοιχη νομοθεσία κατά των βασανιστήριων, που το ακούσαμε και προηγουμένως ε, και συζήτηση με την Υπουργό, την κυρία Πλούμεν. Η πρώτη συνεδρία του Λόγου έγινε το Δεκέμβριο με τη Λουξεμβουριανή τότε Προεδρία, όπου είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων να δούμε, να βολιδοσκοπήσουμε ο καθένα τι θέσει του άλλου και ιδιαίτερα κάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει, εκλήθη ε, μάλλον, να κάνει προτάσεις συμβαστικές και ελπίζω γρήγορα να έρθουμε σε ένα αίσιο πέρα και σε καλό δρόμο. Και το δεύτερο είναι τα περίφημα ρηκτά από τις εμπόλεμες περιοχές και η πρώτη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου θα γίνει την άλλη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Αφού το Συμβούλιο επιτέλου στις 18 Δεκεμβρίου έδωσε εντολή για την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Οπότε θα δείξει. Την άλλη Δευτέρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσει. Ούτε καθόλου εύκολε θα είναι, διότι οι θέσει ε, απέχουν πραγματικά πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη εκ των προτέρων έχει κάνει κάποιες προτάσει. Η κυρία Κέλλερ ε, απεχώρησε από τη διαπραγματευτική ομάδα και την αντικαθιστά κυρία Σαρχεντίνη. Πάμε στο 12 λοιπόν που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γιώργ Βούτκε, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα. Και ενώψει και των συζητήσεων που επίκυνται, και της απόφασης για την απονομή του καθεστώτος οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που θα έχουμε στη συνέχεια. Και λόγω του γεγονότος ότι είναι 1.800 και πλέον οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, 1.800. Και ε, το θέμα αυτό τους αφορά το καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας αγοράς. Οπότε ε, έχει ενδιαφέρον να ανταλλάξουμε απόψεις με το ε, επιμελητήριο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βούτκε και μετά στον κύριο Βίνκλερ, τον μόνιμο εισηγητή μας. Παρακαλώ κύριε Βούτκε, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κύριε κύριε, ευχαριστώ πολύ. Α, μισό λεπτό. Ε, πόσο χρόνο έχω. 10-15 λεπτά, λιγότερο 10 λεπτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Ήμουν εδώ πέρσι, Ιανουάριο. Βέβαια, στην Κίνα έγιναν φοβερά και τρομερά πράγματα το τελευταίο χρόνο. Πέρσι τον Ιούνιο ξεκινήσαμε την έκθεση οικονομικής εμπιστοσύνης και οι επιχειρήσεις μας έλεγαν ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα όχι μόνο λόγω της επιβράδυνσης της κινέζικης οικονομίας, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ορισμένοι περίμεναν, αλλά και διότι το κανονιστικό περιβάλλον δεν ήταν τόσο ελκυστικό. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιδρούν, κάνουν ότι μπορούν, αντιδρούν, απολύουν κόσμο, κλείνουν μερικές παραγωγικές εγκαταστάσεις, αλλά δεν φεύγουν από την Κίνα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλη Κίνα δεν υπάρχει. Η Κίνα παραμένει πολύ ενδιαφέρουσα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εκεί επενδύουν και ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Τώρα, η μετοπική άνεμη, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει και τις επενδύσεις. Εκεί βλέπετε σαφώς ότι οι κινέζικες επενδύσεις στην Ευρώπη αυξάνονται κατά πολύ θεματικά. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, οι κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη ήταν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση πάνω από 36%, ενώ οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Κίνα μειώθηκαν κατά περίπου 23% σε κάτι λιγότερο από 10 δισεκατομμύρια. Οι Κινέζοι λοιπόν έχουν επενδύσει τα διπλάσια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε επενδύσει εμείς στην Κίνα. Μας αρέσει αυτό, το καλωσορίζουμε, αλλά ως Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά διαρωτώμεθα γιατί εμείς δεν μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο. Υπάρχουν φυσικά τα κανονιστικά εμπόδια και οι άλλοι παράγοντες που ανέφερα. Υπάρχουν 800 σημεία στα οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί η Κίνα και να βελτιώσει τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας με την Ευρώπη. Το καλοκαίρι βεβαίω ήταν αποκαλυπτικό για πολλούς λόγω της ε, εξέλιξης στα κινέζικα χρηματιστήρια στα μέσα του Ιουνίου ο δείκτης από 2.000 ανέβηκε στο 5.000, ε, εκτοξεύτηκε στα ουράνια σε σχέση με το 2014 και μετά άρχισε να πέφτει. Και δεν έχουμε καταλάβει ακόμη γιατί επέτρεψε τη φούσκα αυτή η κινέζικη κυβέρνηση. Γιατί δημιούργησε πολλά προβλήματα με τα οποία παλεύει ακόμη η Κίνα. Η κινέζικη αγορά ουσιαστικά έχει αποκοπεί από την πραγματική οικονομία η Κίνα αυξανόταν διαρκώς με 10% το χρόνο. Τα χρηματιστήρια ακολούθησαν, όμως ε, το 2015 αφού έφτασε στα, ο δείκτης στο 5.000 ε, καταπαραθρώθηκε στο 3.000, στις 3.000 μονάδες και μετά αναγκάστηκε η κινησική κυβέρνηση να αρχίσει να παρεμβαίνει, να σταματάει το short selling, να απαγορεύει το short selling, να κλείνει εταιρείε που να αποσύρει εταιρείε που δεν επένδυναν από το χρηματιστήριο ή να πετύχει κάποια σταθερότητα. Στις 4 Ιανουαρίου είχαμε όμως άλλη θεμερική πτώση του χρηματιστήριου. Ε, τώρα κάποιες μετοχές που είχαν αφαιρεθεί από το δίκτυο τον Αύγουστο θα επανέλθουν, άρα δεν περιμένουμε ο δίκτυος να τα πάει πολύ καλά. Μεγάλη λοιπόν ε, αβεβαιότητα, αλλά και μεγάλη βεβαιότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Δείτε τον DAX, η Σανχάη και ο Σανχάν ε, είναι δείκτες οι οποίοι μόνο ανησυχίες ε, γεννούν στην Ευρώπη. Τώρα η θέση μας που εκδώσαμε τον Σεπτέμβριο περίχεται εξής στοιχεία. Το 2014 εξετάσαμε τις υποσχέσεις της κοινωνικής κυβέρνησης από την προηγούμενη χρονιά Ήταν ε, η πρώτη φορά που η κινησική κυβέρνηση είχε καταρτήσει έναν χάρτη πορείας, τα στιβαρό θα έλεγα. Και γι' αυτό λοιπόν από πέρσι τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισαμε να συμμετοδοτούμε τις προβλέψεις με κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο, άρχισαμε να στέλνουμε τα πρώτα αρνητικά μηνύματα. Μόνο το 20% πάντως προβλέπει ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Το 70% περιμένει λίγο πολύ τα ίδια. Ε, κρίμα διότι ο χάρτης αυτό πορείας δείχνει ότι η κινέζικη κυβέρνηση ποντάρει στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία. Προσπαθεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Από τότε που τα είπαμε πέρσι, το κινέζικο νομίσμα συμμετέχει στο στα στα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Αυτό έχει μεγάλη συμβολική σημασία. Έτσι η Κίνα διεθνοποίησε το Ρεμίμπι. Η ευελιξία των επιτοκίων αυξήθηκε και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν μια πραγματική μεταρρύθμιση. Γίνεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας να έρθει πιο κοντά στο ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Φέτο το Ρεμίμπι θα είναι το τρίτο αποθεματικό νομίζω μετά το δολάριο και το ευρώ. Επίσης, η κινέζικη οικονομία ανοίγεται περισσότερο στις παγκόσμιες αγορές, κάτι το οποίο μεταφέρει όμως ε, στην Κίνα την αβεβαιότητα που παρατηρήθηκε στα χρηματιστήρια τον Ιανουάριο. Όπως είπα, ο δείκτης έχει πέσει κάτω από 3.000 και φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός θα πέσει και άλλο δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχουν περάσει ακόμα τα χειρότερα. Τα άλλα που σημειώσαμε ω επιχειρήσει είναι ότι η Ευρώπη συνεργάζεται πλέον με την ασιατική επενδυτική ε, τράπεζα, μια τράπεζα που ιδρύθηκε από την Κίνα, είναι μια αναπτυξιακή τράπεζα η οποία κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμμετάσχουν και στα, στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί είπαμε όχι. Έχει πάντως μεγάλη σημασία ότι κάποιοι Ευρωπαίοι βρίσκονται στο ΔΣ της τράπεζας αυτής. Έτσι δυσφαλίζουμε ότι οι όροι των προμηθειών της κινέζικης κυβέρνησης θα είναι πιο διεθνείς και όχι μόνο κινέζικοι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η τράπεζα αυτή θα ακολουθήσει τις διεθνείς πρακτικές και όχι τις κινέζικες. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν πραγματικά για, τις, για την ανάπτυξη των υποδομών. Αν κατάλαβα καλά, το πρώτο μεγάλο έργο που θα χρηματοδοτήσει αυτή η Κινέζικη Αναπτυξιακή Τράπεζα θα γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μετά, πέρα από τον παραδοσιακό δρόμο του μεταξιού, έχουμε και το θαλάσσι, τους θαλασσιούς δρόμους. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα περνάει από το Καζακστάν και είναι προτεραιότητα για τον Κινέζο Πρόεδρο. Περιμένουμε πάντω να δούμε που, τι θα κάνουν. Δύο χρόνια περιμένουμε. Είχαμε εξαγγελίε τη μία μετά από την άλλη. Περιμέναμε πολλά από την απελευθέρωση του τομέα των ε, υπηρεσιών. Ισμάτιν όμως. Δηλαδή από συμβολισμό και εξαγγελίε μια χαρά πάνε οι Κινέζοι τον τελευταίο καιρό, το μάθαμε. Ε, αλλά δυστυχώ απογοητευόμαστε. Κάτι μάθαμε πάντω. Είστε στις 22 Φεβρουαρίου στο Πεκίνο θα ανακοινώσουμε έκθεσή μα σχετικά με τους βασικούς κλάδους του χάλιβα, του τσιμέντου. Εκεί δείχνουμε ότι υπάρχει υπερβάλλους παραγωγή, υπερβάλλον δυναμικό, πάνω από αυτά τα οποία ζητάει η αγορά. Ειδικά κρίση του χάλιβα αφορά πλέον και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά λέμε αυτά που κάναμε, λέμε αυτά που λέμε, που κάναμε το 2009. Πρόκειται για μια μελέτη που βέβαια δύσκολα δεν διαβάζει κανείς. Οι Κινέζοι πάντως προτιμούν την, ε, το περιβάλλον δυναμικό, την υπερβολική παραγωγική δυναμικότητα γιατί έτσι πέφτουν οι τιμές. Εμείς ανησυχούμε πάντως, διότι το κινέζικο νομίσμα είναι υποπίεση, διαραίουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα αυτή τη στιγμή από την Κίνα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η προσφορά, αλλά και το θέμα του νομίσματος. Οι βασικές λοιπόν ανησυχίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το χρέος της κινέζικης οικονομίας, που δεν είναι μόνο υψηλό σε απόλυτε τιμές, αλλά έχουμε και ένα νούμερο το. Από το 140 έχουμε πάει στο 240% του κινέζικου ΑΕΠ, κατά τη Μακένση. Είναι ένα σεισμό αύξηση που δεν έχουμε δει πουθενά αλλού. Φυσικά η κινέζικη οικονομία διαφέρει από όλε τι άλλε. Παρ' όλα αυτά ανησυχούμε. Το χρέο αυτό πρέπει να εξυπηρετηθεί. Μειώνονται οι χρηματοοικονομικέ ε, ροέ που βεβαίω έχουν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση τη οικονομία. Όταν τα χρήματα λοιπόν πηγαίνουν στην αποπληρωμή των δανείων και όχι στην πραγματική οικονομία. Το 2016 λοιπόν πιστεύω ότι στην Κίνα θα είναι δυστυχώ ε, η χρονιά με τα άσχημα νέα λόγω τη επιβράδυνση τη οικονομία, λόγω τη φυγή κεφαλαίων, λόγω των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει το Ρεμίμπι, θα υποτιμηθεί κατά πάνω από 5% και λόγω του διεθνού περιβάλλοντο αβεβαιότητα. Εκεί θεωρούμε ότι η Κίνα πρέπει κάτι να κάνει για να αναστρέψει την πορεία αυτή. Πού θα μπορούσαμε να έχουμε καλά νέα. Σε ποιου τομεί. Πρώτον στην επενδυτική συμφωνία που διαπραγματεύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την Κίνα. Οι Κινέζοι, όπως είπα, έχουν διπλάσεις επενδύσει στην Ευρώπη, υποτιμήσει στην Κίνα. Αυτό είναι ένα. Ε, Μά όμω δεν μα ενδιαφέρει η προστασία των επενδύσεων τόσο πολύ όσο η πρόσβαση στην αγορά. Με τον Επίτροπο, λοιπόν, τι επόμενε μέρε θα προσπαθήσουμε και θα πούμε στου Κινέζου μην βιάζεστε. Το θέμα είναι οι συμβολισμοί να έχουν και σημασία, να έχουν περιεχόμενο συγκεκριμένο. Αυτά εν ώψη τη νέα συμφωνία, η οποία πρέπει να παρέχει πρόσβαση στην αγορά. Θέλουμε λοιπόν μια καλή συμφωνία παρά ταχύτερα μια κακή συμφωνία. Αυτό είναι ζωτική σημασία για μας. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσουμε φέτος ή αρχές του 2017. Οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή με τους Κινέζους επίσης. Θα τους προφτάσουμε όμως. Από τα δεδομένα των επενδύσεων βλέπουμε ότι οι Κινέζοι βλέπουν πολύ πιο ευμενώς τους ε, Ευρωπαίους παρά τους Αμερικανούς. Υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις 50 δισεκατομμυρίων. Όταν ήμουν εδώ πέρσι, πριν από ένα χρόνο, είχα, ρωτήσει, είχα ζητήσει μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο πράγματα. Είχα, πει, ό,τι κάνει το Αμερικανικό Κογκρέσο, κάντε το κι εσεί παρακαλώ. Ε, μια ετήσια έκθεση μια έκθεση για τι εμπορικέ σχέσει με την Κίνα. Για περισσότερη διαφάνεια, για το που βρισκόμαστε, τι προβλήματα υπάρχουν και πού πηγαίνουμε. Ύστερα ζήτησα την υποστήριξή σα την ε, Συμφωνία για τι Επενδύσει και για περισσότερη διαφάνεια με στόχο τον περιορισμό των περιορισμών. Και τέλος, αυτό που σας ενδιαφέρει όλους πολύ κύριε Πρόεδρε, είναι ο χαρακτηρισμός οικονομία της αγοράς. Κοιτάξτε, ούτε η Κίνα, ούτε η Ρωσία, ούτε η Βιετνάμ φυσικά πληρούν αυτόν τον ορισμό. Το θέμα είναι ότι είχε δοθεί υπόσχεση το 2001. Το <laughs> τραγικό σε αυτήν την συζήτηση, το οποίο δεν το λένε οι δημοσιογράφοι, είναι ότι ο Πρωθυπουργό Τζου το 2001 ήθελε 15 χρόνια, έχει ζητήσει 15 χρόνια προσαρμογή πριν ε, γίνει, έλεγε, η Κίνα οικονομία αγοράς. Από αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν πραγματικά δυνάμεις αγοράς όπως καταλαβαίνουμε στην αγορά και αυτό είναι κρίμα για τη χώρα. Η Κίνα έχει να κερδίσει, πιστεύω, εάν προσπαθούσε πραγματικά να γίνει η οικονομία της αγοράς. Ε, δεν κατηγορώ αυτήν την κυβέρνηση της Κίνας γιατί και η προηγούμενη είχε πετύχει η αύξηση της οικονομίας 10% το χρόνο και δεν γιατί πρέπει να αλλάξει κάτι. Τώρα, στην τρίτη ολομέλεια, έγινε λόγος για τις, οικονομ... για τις δυνάμεις της αγοράς και ελπίζω ότι δεν θα τα παρατήσουν στη μέση και θα συνεχίσουν να προωθούν τις αλλαγές που θα κάνουν τη χώρα πραγματικά μια οικονομία της αγοράς. Ευχαριστώ κύριο Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς για αυτή την έκθεση και την ενημέρωση κύριε Βούτκε. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει γιατί αφορά όχι απλώς την Κίνα αλλά και άλλες χώρες ε, της ίδιας γεωγραφικής ζώνη Ίσως είναι η χρονιά με τις άσχημες ειδήσει αυτή. Οι πιθανότητες για καλές ειδήσει θα προέλθουν από επενδυτικές συμφωνίες όπως είπατε και εσείς κύριε Βούτκε οι οποίες μπορεί να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2016 ή στις αρχές του 2017. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι αίσθηση έχετε, τι μηνύματα λαμβάνετε, γιατί εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε στις Βρυξέλλες είναι ότι υπάρχει κάποιο είδους ε, διαπλοκή, για να μην πω ασχετισμός, η αιρεσιμότητα, Δηλαδή η δική μας στάση για το αν θα αποδώσουμε καθεστώς οικονομίας της αγοράς θα καθορίσει το αν θα υπάρξει διάθεση για πρόοδο από την κινέζικη πλευρά. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση. Συμμερίζεστε αυτή την αίσθηση κι εσείς. Και η δεύτερη μου ερώτηση μιλήσατε για το μία ε, γεωγραφική ζώνη, ένας δρόμος. One belt, one road. Ε, συζητά εντατικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Κίνα το θέμα αυτό και ε, στην παρουσίασή σας στο αμέσως επόμενο σημείο περάσατε στην ε, υπέρμετρη ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας και αναφέρατε και κάποιους τομείς Τι σχετισμό βρίσκεται κύριε Βούτκε μεταξύ αυτής της υπερδυνατότητας ε, του, του υπερβολικού δυναμικού που διαθέτουν τα κοινωνικά υπουργεία και την προθυμία τους να συνεργαστούν επαρκώς με τους Ευρωπαίους εταίρους. εταίρους. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Τρεις ζητούν το λόγο τώρα. Είμαι πρώτη και μετά γιοτήτη. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας και τα λόγια σας. Θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, Ε, οι Κινέζοι, ειδικοί αναλυτές, ε, πανεπιστημιακοί και τα λοιπά έχουν κάνει καμιά ανάλυση για το πώς υλοποιείται η Συμφωνία Πρόσβασης στον ΠΟΕ από πλευράς Κίνας. Έχει γίνει καμιά μελέτη, καμιά αξιολόγηση σχετικά. Δεύτερον, τι γίνεται σήμερα με τις απομιμήσεις και τα προϊόντα μαϊμού βασικά. Ε, τι γίνεται με τα κινέζικα αυτά προϊόντα που είναι απομιμήσεις και παραποίηση προϊόντων και τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τρίτον, είπατε κάτι με το οποίο συμφωνώ και φαντάζομαι όλοι γνωρίζουν. Η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς, μόνο. Είναι ε, κεντρικά σχεδιαζόμενη οικονομία και αυτό ε, από χέρι είναι ασύμβατο με την οικονομία της αγοράς. Αλλά ας πούμε, στην υποτιθέμενη περίπτωση που η Κίνα λάβει το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, πώς αυτό θα ε, επηρεάζει τον υπολογισμό του dumping. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, το ψάχνει ο επιχειρηματικό κόσμος αυτό. Υπάρχει καμιά μέθοδος για να μπορέσουμε να μετράμε το dumping και να αντιμετωπίσουμε και ενδεχόμενα τέτοια και ε, αθέμητο ανταγωνισμό ενδεχομένω. Ευχαριστώ. Τώρα η Τζούτ. Δεν κατάλαβα την πρώτη ερώτηση γιατί δεν είχα βρει τη διερμηνία. Ναι, να την επαναλάβω. Η Κίνα δεσμεύτηκε, όπως είπατε κι εσείς, και τα ξέρουμε όλοι, για να μπει στον ΠΟΕ. Δεσμεύτηκε ότι θα κάνει χι πράγματα ε, για την ίδια την πρόσβασή τη. Και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν προσχώρησε, έκτοτε έχουν γίνει μελέτε από πλευρά κινέζικων αρχών, εμπειρογνωμών, αναλυτών, οι ίδιοι Κινέζοι το έχουν μετρήσει, τα πανεπιστήμια έχουν αξιολογήσει το βαθμό συμμόρφωση τη κίνα προ τι υποχρεώσει που αναλάμβανε όταν υπέγραψε τη Συμφωνία προσχώρηση ένταξή τη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Um, Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γούτκε για αυτή την αρκετά ανησυχητική παρουσίαση του πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Θα μπορούσε να το δει κανείς και από τις σελίδες περί επιχειρήσεων ε, στις εφημερίδες μας. Δεν προβλέπονται πολύ καλά τα νέα για τη διεθνή οικονομία. Απλώς μια γρήγορη ερώτηση. Είπατε ότι το φως στην άκρη του τούνελ ίσως να είναι αυτή η διμερής επενδυτική συνθήκη και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα έφτασαν σε συμφωνία για το πεδίο μιας τέτοιας ενδεχόμενης μελλοντικής διμερούς ε, συμφωνίας για, την, για τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα υπάρχει ένα υψηλό και ισόρροπο επίπεδο προστασία για του επενδυτέ και τι επενδύσει του, εφόσον η συμφωνία εγκριθεί. Ε, δεν είναι ακριβώς αυτή η ερώτησή μου, αλλά είναι σαφέ ότι η ευρωπαϊκή πλευρά και η κινέζικη θέλουν να υπάρξει ένας μηχανισμός επίλυση των διαφορών επενδυτικού κράτου στι περιπτώσει αυτέ και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συνθήκη. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε μπορεί να έχουν να αντιμετωπίσουν γεωπολιτικέ πιέσει εφόσον μετατοπιστούν στην Κίνα και δεν έχουμε αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτέ οι εταιρείε βάσει των διμερών συμφωνιών που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών και Κίνας, γιατί σχεδόν κάθε κράτος μέλος έχει διμερή ε, επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι εταιρείε αυτέ έχουν ε, καταφύγει στον μηχανισμό επίλυση των ε, διαφορών. Μόνο δύο υποθέσει λέει βάσει δεδομένων ότι υπήρξαν με προσφυγή κατά τη Κίνα από το 1992 και σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει φόβο για αντίπεινα από την κινέζικη κυβέρνηση ή καμία εταιρεία δεν είχε πρόβλημα ή δεν το έθεσε. Σε αυτήν λοιπόν την υποθετική, σε αυτό το επιθετικό σενάριο, ε, εάν ο μηχανισμός ISDS υπάρχει στη Δημερή Συμφωνία, θα κάνει κάποια διαφορά για τις εταιρείε ή όχι. Ή μήπω η όλη πολιτική κατάσταση γίνει πολύ περίπλοκη και τελικά δεν ε, καταλήξουμε σε κάποια λύση. Ευχαριστούμε κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ. Τα περισσότερα σχόλιά μου έχουν καλυφθεί από τους συναδέλφους, αλλά θα ήθελα να ακούσω για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κίνα. Τι άποψη έχετε για την δική τους θέση ως προς την απόδοση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Και επίσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαγράψει στην Κίνα τον κατάλογο ε, των δασμολογικών ε, δυσκολιών. Επίσης θα υπάρξει διάλογος για την περίπτωση αυτή της οικονομίας της αγοράς από το ΠΟΕ ή ίσως προβλεφθούν διμερείς κυρώσεις. Θα, μας δείξει, θα μπορούσατε να μας πείτε τι γεύση και τι εικόνα έχουν για το θέμα αυτό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιτόπου. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει τίποτα. Όχι. Α, θέλει. Παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Να πω απλώς ότι το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο εμπορικό επιμελητήριο στην Κίνα είναι πολύ σημαντικό συνομιλητή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την DigiTrade ιδίω. Έχει κάνει τεράστιο έργο περνώντα πληροφορίε ε, για το θέμα που μα ενδιέφερε και για να καθορίσουμε τη στάση μα και το σχετικό έγγραφο και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τι εταιρείε μα στην Κίνα. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα την φύση των προβλημάτων και μπορούμε να παρέμβουμε όταν έχουμε συζητήσει με του ε, Κινέζου εταίρου μα. Οι ομολόγους ή να διευκολύνουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείε για τις, για τις δουλειές τους, την στρατηριότητες τους στην Κίνα. Το έγγραφο αυτό, Πρόεδρε, σα έχει υποβληθεί γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Μετρά καταγράφει μάλλον τα μέτρα τη κινέζικη κυβέρνηση και τι προθέσει τη να μεταρρυθμίσει τον τομέα τη οικονομία. Μεταρρυθμίσει απαραίτητε όχι μόνο για την, για την Κίνα, αλλά και για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε και του υπόλοιπου εμπορευομένου στην κινέζικη επικράτεια. Γι' αυτό στηρίζουμε το έγγραφο και νομίζω ότι είναι μια κοινή συνθαρρυντική για όλου μα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε την Κίνα, να μην ε, εγκαταλείψει τι προσπάθειε για μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα που έχουμε, όπω το υπερβολικό δυναμικό ή τα προβλήματα διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Βούτκε τώρα. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Το θέμα του πώς συνδέεται ο χαρακτηρισμός οικονομία της αγοράς με τις συμφωνίες περί επενδύσεων. Πω, οι Κινέζοι συνομιλητές μας δεν το έχουν θέσει έτσι ποτέ ότι αν δεν υπογράψετε τις συμφωνίες θα υπάρχουν επιπτώσεις τις επενδύσεις. Νομίζω ότι πιστεύουν ότι έχουν οικονομία της αγοράς. Το είχαν υποσχεθεί το 2001 και νομίζω ότι σιγά σιγά έγινε. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι να φτάσουν στον τελικό στόχο πάντως, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι τις επενδυτικές συμφωνίες τις βλέπουν ως ένα βήμα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των κινέζικων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Οπότε από όσο έχω μιλήσει μαζί του τουλάχιστον δεν βλέπω κάποια σύνδεση μεταξύ των δύο ε, δεν ισχύει το ότι αν δεν υπογράψετε τη συμφωνία δεν υπάρχει ξεχάσετε τι επενδύσει. όχι, Τώρα, στην πράξη βεβαίω υπάρχει κάποια σχέση με το θέμα τη περιβάλλουσας δυναμικότητα και το είχε πει ένας Κινέζος αξιωματούχο πρώην υφυπουργό, ο οποίο είπε ότι η όλη προσπάθεια είναι να μην χρειαστεί να πετάξουμε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αλουμινίου ή χάλιβα. Όμως οι ποσότητες είναι τεράστιες. Που δεν υπάρχει τρόπος να απορροφηθούν αυτές οι ποσότητες από το Καζακστάν ή το Κυριστάν ή δεν ξέρω που αλλού. Είναι απλώς αδύνατο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Για να πούμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και δεν ξέρω και κατά πόσον οι χώρες αυτές έχουν και όρεξη να απορροφήσουν τόσο τεράστιες ποσότητες. Τι θα, πόσους σταθμούς θα χτίσουν σιδηροδρομικούς η παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι η λύση. Το One Belt One Road είναι πάντως ένα όραμα το οποίο δεν νομίζω ότι στηρίζεται στην πράξη ρεαλιστικά. Η περιβάλλουσα δυναμικότητα, όπως θα λέει η μελέτη μας, μπορεί να εξελιχθεί, να αμβλυνθεί μόνο με κάποια ουσιαστική αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και αλλού. Κάναμε νέα έρευνες στην ηλιακή ενέργεια, στη χημική βιομηχανία, όχι μόνο στο χάριβα και το αλουμίνιο. Έχουμε θεματικές τέτοιε έρευνες που με χαρά θα στείλω στον πρόεδρο για να τις διαβάσετε. Αν υπάρχουν τώρα μελέτες από κινέζικε αρχέ, ναι υπάρχουν τέτοιε μελέτε και πρέπει να σας πω ότι πληρούν τα κριτήρια του, του ΠΟΕ είναι ότι καλύτερο έχει η Κίνα να επιδείξει κάποιος βεβαίως, ξέρετε, είναι 400 σελίδες, εν πάση περιπτώσει το... η ουσία είναι ίδια, το σελίδων. Ξεκίνησαν μάλιστα να μελετούν και να μελετούμε και εμείς ε, πόσα χάνουμε τελικά ως Ευρώπη λόγω έλλειψη πρόσβαση στην αγορά. Η απάντηση ήταν 70 δι. 70 Το οποίο σημαίνει ότι πολλέ θέσει εργασίας κινδυνεύουν λόγω ακριβώ της ε, δυσκολίας πρόσβαση στην κινέζικη αγορά. Όσον αφορά τώρα τα κλειψίτυπα, ε, από το πάρα πολύ κακό η κατάσταση είναι λίγο, λιγότερο κακή. Δυστυχώς από τα κλειψίτυπα το 80% μπαίνει στην Ευρώπη είναι από την Κίνα και το Χονγκ πρόβλημα υπάρχει, ακόμα και σήμερα. Αλλά δεν στοχεύει μόνο την Ευρώπη. Εμείς είμαστε μικροί παίκτες, θα έλεγα, 95% των περιπτώσεων στην Κίνα στο δικαστήριο για τα πνευματικά δικαιώματα και τις ε, αφορά Κινέζους εναντίον Κινέζων αυτοί που φέρνουν κατά κύριο λόγο γιατί και οι Κινέζοι πρέπει να προστρεφθούν Φυσικά εμείς σίγουρα χάνουμε κάθε φορά που εξάγουν τέτοια προϊόντα μαϊμού οι Κινέζοι. Ε, Βελτιώνουν οι Κινέζοι, αλλά σίγουρα στην εφαρμογή έχουν καθυστερήσει πολύ. Ωραία, σε μια οικονομία που δεν είναι οικονομία αγορά, πώ να προηγήσει κανεί τα ποσοστά dumping. Α το πατήσει κομισιόν, μάλλον ξέρουν καλύτερα, αλλά αν δείτε τι εισαγωγέ από χώρες που είναι οικονομίες της αγοράς, ε, εκεί δεν ξέρω την υπολογίσει κανεί. Το θέμα είναι πόσε περιπτώσει επιδοτήσεων έχουμε. Αλλά εκείνα είπα δεν είναι οικονομία αγορά. Άρα ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Και έχουν και ανταγωνισμό από παρόμοιε χώρε. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Πώ μπορούμε να υπολογίσουμε δηλαδή το ποσοστό του εφαρμοζόμενου dumping για την Σύμφωνη Επενδύσεων είναι παράξενο. Όλη την ζητούμε, αλλά ποτέ δεν τη χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, αισθανόμαστε ασφάλεια με αυτή τη συμφωνία, αλλά όπως είπατε και εσείς, τελικά δεν έπαιξε και ρόλο στις δουλειές μας στην Κίνα. Οι εταιρείε πάντως φοβούνται και σήμερα τα αντίπεινα, δηλαδή αν κυνηγεί στα δικαστήρια την κινέζικη κυβέρνηση, ξέχνα την κινέζικη αγορά. Ξέρω χώρες και επιχειρήσεις που το εξετάζουν σοβαρά να στραφούν δικαστικά κατά υπουργείων, οργανισμών του κοινωνικού δημοσίου κλπ. Το παράτησαν όμως γιατί ε, δεν ε, θέλεις να βρεθείς αντιμέτωπος ε, με τα μεγαθύρια. Οι μεγάλες επιχειρήσεις πάντως έχουν τον τρόπο τους να λύνουν, να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, διότι έχουν πρόσβαση στα, στα υψηλά κλιμάκια Ξέρω μια ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία η οποία ήταν έτοιμη πραγματικά να πάει στη Βηρησία ή να κυνηγήσει στη δικαστήρια τους Κινέζους. Τελικά βρήκαν ε, λύση μέσω υψηλά ειστάμενου στη Μόσχα. Για τις μεσαίες όμως, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Είναι λίγο ακαδημαϊκή η συζήτηση, αλλά να σας πω στην επιχειρηματική κοινότητα ε, η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι Καλύτερα είναι με συμφωνία παραχώρηση. Το θέμα είναι θα την χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Η πράξη δείχνει ότι μάλλον όχι. Όσον αφορά τώρα τα αντίπεινα, ότι αν δεν ε, πάρουν το χαρακτηρισμό η κοινωνία τη αγορά, τι θα κάνουμε τι επενδύσει. Αυτό δεν ε, είναι ψηλά στην προτεραιότητα, πιστεύω, των συνομιλητών μου στο Πεκίνο, διότι απλούστερα δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Δηλαδή, ε, δεν εξάγουμε στην Κίνα, ίσως που είχαμε περιπτώσεις dumping κατά της Ευρώπης, η Business Europe ανησυχεί περισσότερο για τις εξαγωγές των Κινέζων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχουν κάποιες ενώσει. Το θέμα της υπερβάλλουσας δυναμικότητας μας ανησυχεί. Το αν θα προβεί σε αντίπεινα λοιπόν η Κίνα, αν δεν πάρει την, το χαρακτηρισμό οικονομία τη αγορά, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν ποτέ στη Γενέβη για να κινηθούν νομικά. Θα τιμωρήσουν τώρα αλλιώ κάποιε χώρε το έχουν κάνει στο παρελθόν. α πούμε η Νορβηγία ε, μπήκε στο ψυγείο για πολύ καιρό για πολιτικού λόγου πριν από μερικά χρόνια. Όμω θεωρώ ότι η Κίνα το 2016 δεν θα πάει και πολύ καλά έχουν την προεδρία του G20. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα το αφήσουν να πάει έτσι προς τα κάτω το πράγμα ή θα διευκολύνουν ε, τις εξελίξεις. Αυτά. Ε, κλείνω λέγοντας ότι παραμένω αισιόδοξο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε και πάρα πολύ κατατοπιστικά. Πώς αλλιώς να ήταν άλλος. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συντονιστέ, ακολουθεί αμέσω η συνεδρίασή μας, που σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι να πάτε στο καλό. Και πάρα πολύ γρήγορα, αν μπορείτε.